Ε, συνθήκες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό αποτελεί και τη μοναδική νομική δυνατότητα για να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες. Δεν προβλέπεται κάτι άλλο. Είναι λοιπόν ουσιώδης, ουσιώδης σημασία. Γιατί θέλουμε να τηρούμε προφανώς ε, τα κριτήρια τα νομικά σε ό,τι αφορά την τις δραστηριότητε των υπηρεσιών μας σε ένα τρίτο κράτος. Η σύναψη λοιπόν ε, των ε, νομικά δεσμευτικών ε, τέτοιων συμφωνιών αντικαθιστά τα άτυπα της άπειτες συμφωνίες και ουσιαστικά θα προωθήσει την διαφάνεια και την άσκηση δημοκρατικού ελέγχου. Στις συμφωνίες λοιπόν αυτές ότι αφορά τη Σερβία και το Μαυροβούνιο ουσιαστικά ορίζεται η έκταση των επιχειρήσεων, η, τα καθήκοντα και υποχρεώσεις των απεσταλμένων ομάδων. Και θα θέλαμε να τονίσουμε ιδιαίτερως το άρθρο 9 σε ό,τι αφορά τι συμφωνίες αυτές, το οποίο ορίζει τις διατάξεις για την διατήρηση των βασικών δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων, στα οποία προφανώ έχουν δεσμευτεί. Οι βασικές ελευθερίες, λοιπόν, μεταξύ των οποίων και η πρόσβαση στο άσυλο, η αξιοπρέπεια, η ανθρώπινη, η αποφυγή εξετελιστικών καταστάσεων σε ό,τι αφορά επίσης τα δικαίωμα μη επιστροφών και το θέμα των συλλογικών επιστροφών, τα δικαιώματα των παιδιών και το δικαίωμα της, ε, του σεβασμού τη ιδιωτική σφαίρα και τη οικογενειακή ζωή. Επίση, η αρχή τη μη διακριτική μεταχείριση. Τα θεμελιώδη λοιπόν δικαιώματα είναι κατεξοχήν ευαίσθητα ζητήματα επί των οποίων θα πρέπει να εξκύψουμε ως ευρωβουλευτές και θα πρέπει λοιπόν όλοι οι παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεσμεύονται για την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και κυρίως σε ό,τι αφορά την κατάρτιση και την εκπαίδευση των υπαλλήλων θα πρέπει να δοθεί έμφαση εδώ γιατί υπήρχαν περιστατικά σε ό,τι αφορά την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων Και πριν από την έναρξη λοιπόν των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να κοιτάξουμε ε, πώς έχει κατάσταση στο κράτος δικαίου των κρατών αυτών, των τρίτων κρατών αυτών και όλα αυτά θα πρέπει να διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να γίνει λοιπόν μια σωστή αξιολόγηση των συμφωνιών θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, απόλυτη διαφάνεια. Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Εξωτερική Υπηρεσία εγκαίρως να υποβάλουν εκθέσει για τις δραστηριότητε τους στις εκάστοτε χώρε. Και σύμφωνα με τον κανονισμό για τις εξωτερικές υπηρεσίες υπάρχει και υποχρέωση για συνεργασία με κράτη-μέλη τρίτα, με τρίτα κράτη, με τρίτα κράτη συγγνώμη, σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις αυτές τις ε, διαδικασίες και ενεργείες. Και συγκρίνουμε Συγκρίνοντα τι συμφωνίε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διαφορετική διατύπωση και είναι περίεργο το γεγονός ότι ιδιαίτερα στο αφορά το ειδικό καθεστώς κάποιων κρατών μελών υπάρχει διαφορετική διατύπωση και επίσης η ρήτρα α, ε, μη διακριτικής μεταχείρισης και αυτή έχει διαφορετική διατύπωση. Αυτό οδηγεί σε αβεβαιότητες. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαία διατύπωση όλων των διατάξεων. Τέλος, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτές οι δύο συμφωνίες συνάδουν με το μοντέλο τέτοιων συμφωνίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συστήνω λοιπόν να γίνουν περαιτέρω βήματα προκειμένου να δώσει και το Συμβούλιο την ε, έγκρισή του. Και επίση 21 Ιανουαρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ψηφοφορία στις 28 Ιανουαρίου και στην Ολομέλεια ε, το Μάρτιο. του Μαρτίου. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους και προσβλέπω σε μια επικοδομητική συνεργασία μαζί με όλους σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέγει ο Πρόεδρος. Και τώρα, να δούμε τι έχουν να πούν και οι εισηγητές. Οι σκιώδεις. Από το ΕΛΚ, η κυρία Μέτσολα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλή χρονιά εύχομαι. Ευχαριστώ θερμά την Πετίνα Βόλατ για το έργο τη. σε αυτά τα δύο σχέδια σύστασης για την σύναψη της Συμφωνίας περί με το Μαυροβούνιο και τη Σερβία και κυρίως για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Εκτοφυλακής στην επικράτεια των δύο χωρών. Όπως είπαμε, δεν είναι η πρώτη συμφωνία περί για την οποία δίνουμε σύσταση από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελούν ένα απόσπαστο τμήμα οι συμφωνίε αυτέ του νομικά δεσμευτικού πλαισίου των επιχειρήσεων των οργανισμών όπου αναπτύσσονται μέλη με εκτελεστικέ εξουσίε. Επίση, α μην ξεχνούμε ότι αυτέ οι συμφωνίε περί καθεστώτο προβλέπονται στα πλαίσια του πρώτου κανονισμού, του 2016 δηλαδή, που αντικαταστάθηκε στο μεταξύ από τον κανονισμό του 2019, τον οποίο παρακολούθησα ως εισηγήτρια αρμόδια. Οπότε οι αναθεωρημένες διατάξεις του τελευταίου κανονισμού για τα θέματα αυτά ε, αντα, αντανακλώνται και στα επιχειρησιακά σχέδια αυτών των συμφωνιών περί καθεστώτος. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της ομάδας ΡΙΝΙΟΥ. Ε, ο κ. έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε συγγνώμη. Ε, ευχαριστώ και την εισηγητρία. Θα είμαι εξαιρετικά λακωνικό. Η ομάδα Renew Europe με χαρά θα υποστηρίξει την έκθεση που ουσιαστικά δίνει τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις δύο συμφωνίες περί καθεστώτος. Είμαστε ανέκαθεν ε, υπέρμαχοι του οργανισμού Frontex και υπέρ των νομικά δεσμευτικών διατάξεων σε ένα πλαίσιο που προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις ε, με διαφάνεια και λογοδοσία για τις επιχειρήσεις της του Frontex σε τρίτες χώρες. Γι' αυτό είναι και ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες αυτές οι δύο συμφωνίες. Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους ζητήματα που ανέφερε η συγγήτρια, έχουμε κάποια ίσονο σημασία ζητήματα στις συμφωνίες περί καθεστώτος με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Υπάρχουν αρκετές διαφορές στη διατύπωση σε ό,τι αφορά την ποινική ευθύνη, για παράδειγμα, και για το κατά πόσο ε, τα μέλη του οργανισμού μπορούν να εμφανίζονται ως μάρτυρες σε δίκες στη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Υπάρχουν διαφορές για τα θέματα αυτά στις δύο συμφωνίες, κάτι που είναι παράδοξο και στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε ενιαία διατύπωση σε όλες τις συμφωνίες περί καθεστώτος. Και υπάρχουν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και αποφυγής των διακρίσεων που αναφέρονται αυτό που θα αναμέναμε συνήθως από τέτοιο κείμενο είναι να, έχουν, ε, να έχει ρητή μνήα είτε του ενωσιακού δικαίου είτε των διεθνών συμφωνιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπω το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, για παράδειγμα, ή την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κάτι που δεν βλέπουμε στη συγκεκριμένη συμφωνία. Βέβαια, η διατύπωση είναι καλή και αντιγράφει ουσιαστικά το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Για ζητήματα όμω ασφάλεια δικαίου, και νομική σαφήνεια, καλό θα ήταν να έχουμε ρητήμνια αυτών των κειμένων. Πάντω είναι δευτερεύοντα αυτά τα ζητήματα, όπω σα είπα. Γενικώ ε, χαιρετίζουμε και, την έκθεση, και τι δύο εκθέσει Βόλατ και τι δύο συμφωνίε και με χαρά θα τι υπερψηφίσουμε. Εκ μέρου των Πρασίνων τώρα, ο Ρωμαίο Φραντ είναι ο σκιώδη ηγετή. Δυστυχώ απουσιάζει ο συνάδελφο. Μήπω θα μπορούσα εγώ να πω εκ μέρου των Πρασίνων την άποψή του, ναι. Καλή χρονιά και μπορείτε να τον αντικαταστήσετε. Και εμείς συμφωνούμε με την εισηγήτρια για την ανάγκη διαφάνειας και ομοιόμορφων ρητρών. Και επίσης θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο Frontex επιχειρεί εκτός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας και εφαρμόζει το κοινοτικό κεκτημένο και φυσικά και το χάρτη και συμφωνώ να έχουμε ρητήμνια αυτών των σημείων. Πάντως εκφράζω την ε, ευγνωμοσύνη μου προς την εισηγήτρια για τις διεκθέσεις, οποίες, όπως σας είπα, υποστηρίζουμε. Σας ευχαριστώ εκ μέρους, εκ μέρους του ΡΙΣ ECR. Ο κύριος Στανίσοφ Μπρουτζίνσκι είναι ο σκιώδης εισηγητής, ο κύριος Ποκατσίνη, μια και απουσιάζει ο κύριος Μπρουτζίνσκι. Θα ήθελα απλώ να πω ότι απουσιάζει ο αρμόδιος συνάδελφος, πάντως και η ομάδα συντηρητικών μεταρρυθμιστών συμφωνεί με την εισηγήτρια και το περιεχόμενο των εκθέσεων. Μάλιστα. Η σειρά Ρέγκο για την ΚΟΕ, ούτε και εκείνη. Εσείς αναπληρώνετε. Δεν έχω παρακολουθήσει το θέμα, αλλά μια και δεν είμαστε υπέρ τη επιχείρηση των Frontex σε τρίτε χώρε, εμένουμε σε αυτή τη θέση. Θεωρούμε ότι δεν είναι υπάρχουν ασφαλιστικές δεκλίδες. Ειδικά στην περιοχή αυτή είναι πολύ σημαντικό να τηρούνται, γιατί έχουμε διαπιστώσει σοβαρές παραφιάσεις και του ενωσιακού δικαίου και του διεθνούς δικαίου. Γι' αυτό εμένουμε στη θέση μας κατά, ε, κατά των επιχειρήσεων του Frontex εκτός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Της Επικράτειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, ας ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Όλιβερ Σέιφαρτ. Υπάρχει εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι δεν είναι. Παρακαλώ, κύριε Σέιφαρτ. Ευχαριστώ και καλημέρα σα και καλή χρονιά. Όπω γνωρίζετε, στα μέσα ε, του 2015 η μεταναστευτική κρίση χτύπησε και η οδός των Δυτικών Βαλκανίων ήταν από τις βασικές. Τότε ο Φροντέξ δεν είχε εντολή ε, για να αναπτύξει συνοριοφύλακες ε, σε γειτονικές χώρες. Γι' αυτό και το 2016 όταν ε, συμφωνήθηκε ο κανονισμός για την ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή δόθηκε στο Frontex η δυνατότητα ανάπτυξης ομάδων συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων και στην επικράτεια τρίτων χωρών. Φυσικά μετά από συμφωνία με τις ενδιαφερόμενες χώρες και βάσει αυτής της συμφωνίας περί καθεστώτος. Όπως ανέφερε και η συγκήτρια και στο παρελθόν και πριν τη θέση ισχύ ε, του κανονισμού είχαμε ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με, με όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τις πέντε πριν τη θέση ισχύ του κανονισμού για τον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής. Οπότε ε, με βάση τον κανονισμό 2016 οι συμφωνίες ε, εφαρμόζονται με την πιθανή ανάπτυξη και των ε, συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων της, του Frontex πριν τα τέλη του έτους. Θα δούμε βέβαια κατά στη δυνατό κάτι τέτοιο γιατί θα εξαρτηθεί και από την, πρόοδο, από την που θα σημειώσουμε και με τις πέντε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Για μας πάντως αυτό που ήταν σημαντικό και προχή ήταν να τηρήσουμε την, πρότυπη συμφωνία περί καθεστώτος στο μέτρο φυσικά του δυνατού. Βέβαια, η διαπραγμάτευση με κάθε χώρα ακολούθησε τη δική της δυναμική. Γιατί και τα συμφέροντά τους είναι διαφορετικά και η κατάσταση στις χώρες αυτές ήταν διαφορετική. Αυτό που κατάφερε πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να εφαρμόσει μια οριζόντια προσέγγιση για τα θεμελιώδη στοιχεία, δηλαδή για την ασυλία μόνο για την άσκηση καθήκοντος και την ε, ανάπτυξη ε, των ομάδων της Frontex μόνο στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, βάσει του κανονισμού 2016, κάτι που διαφέρει με την αναθεώρηση του κανονισμού και τον κανονισμό του 2019. Και οι αρμοδιότητες των επιτελείων της Frontex, των ομάδων της Frontex, είναι ίδιες σε όλες τις συμφωνίες. Και οι κανόνες για τις ε, βλάβες και οι, οι για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ίδιες σε όλες τις συμφωνίε. Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναφέρθηκε, υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές στις δύο συμφωνίες. Για παράδειγμα, στη συμφωνία με τη Σερβία, αφενός η Σερβία δεν ήθελε μνήα στον έλεγχο της ταυτότητας, γιατί κάτι τέτοιο ε, δεν αναφέρεται στο σερβικό δίκαιο. Και όπως είπαν και οι σκιώδεις ο Frontex και η Ευρωπαϊκή οι ομάδες ε, τη Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Εκτοφυλακή δεσμεύονται πλήρω από το κοινοτικό κεκτημένο. Οπότε οφείλουν να τηρήσουν και το άρθρο 10 τις οδηγίες ε, για τα χαρακτηριστικά ε, που θα πρέπει να έχει κάποιος για να ζητήσει άσυλο. Κάτι που περιλαμβάνει και την ταυτότητα του φίλου, gender identity σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, νομίζω ότι καλύπτεται από το άρθρο 12 που αναφέρει τις λοιπές διεθνείς υποχρεώσεις. Οπότε υπογραμμίζουμε εδώ ότι όλες οι διεθνείς υποχρεώσεις που φέρουν ήδη τα Δυτικά Βαλκάνια, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων εφαρμόζονται πλήρως όπως η Ευρωπαϊκή η, σύμβαση, ε, η Διεθνή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Θέλουμε και οι πέντε συμφωνίες να καταστούν λειτουργικές μέχρι τα τέλη του έτους. Και φυσικά συμφωνούμε απόλυτα με την εισηγήτρια ότι καλό είναι να κρατούμε μια κοινή προσέγγιση και εναρμονισμένη και στις πέντε συμφωνίες. Θα λάβουμε φυσικά υπόψη και το νέο κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Φυλακή και Ακτοφυλακή που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο και θα αναθεωρήσουμε αντίστοιχα και εναρμονισμένα και τις πέντε συμφωνίες περί καθεστώτος. Και φυσικά θα προσπαθήσουμε ε, να εναρμονίσουμε τις μικρές αυτές διαφορές που παρατηρήσατε στις διάφορες συμφωνίες. Τώρα, κάποιος και ο αναφέρθηκε στη παρουσία των μελών του Frontex ως μαρτύρων σε δίκες. Για τους μάρτυρες λοιπόν, η αλλαγή που έγινε, έγινε μετά από αίτηση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων ε, να καλούνται μάρτυρες και τις εθνικές δίκες. Βέβαια, Παρατηρήσαμε τη συμφωνία περί και προσθέσαμε ένα επιπλέον στοιχείο. Αλλά δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Είναι μια μικρή προσθήκη που ήταν σημαντική για τη συγκεκριμένη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτά και νομίζω ότι σχολίασα όλες τις παρατηρήσεις των σχεδόν εισηγητών και της εισηγητρίας. Μάλιστα, η κυρία Μπόλατ έχει και πάλι το λόγο. Βόλατ. Σα ευχαριστώ, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και του κοιότε για αυτά που σχολίασαν και για τι εξήγησει που μα έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσωπικά θα ήθελα να τονίσω κλείνοντα το εξή ότι θα ήθελα η κοινή αυτή δράση τη υπηρεσία ε, στι χώρε αυτέ ε, βάσει των συμφωνιών καθεστώτο καταρχά να οδηγήσει σε πιο πολύ ασφάλεια και κατά δεύτερον στην τήρηση των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων. Είτε μιλάμε για τέτοια δικαιώματα τα οποία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή από τις συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα αντιδεσμευτικό. Θα πρέπει να ισχύουν και τα δύο αυτά σκέλη σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και επίσης πιστεύουμε ότι θα σημαίνει αυτό μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και μεγαλύτερη υπευθυνότητα στη ε, συνεργασία με τις χώρες αυτές των Δυτικών Βαλκανίων. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν καλύτερη συνεργασία η οποία είναι κάτι που χαιρετίζουμε όλοι και προσβλέπω στις μελλοντικές ε, επικοδομητικές εργασίες και σας ευχαριστώ. Okay. Μάλιστα. Λέει ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. That leads us to the following point in the order of the day. Περνάμε στο επόμενο θέμα, στην ημερήσια διάταξη, το 6. Ερώτηση προς την Κομισιόν για γραπτή απάντηση, 18 Σεπτεμβρίου 2019 για την παράνομη χρήση της βάσης δεδομένων ε, του συστήματος Σέγγεν από τις ε, αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για διάφορα μέλη της ομάδας ΡΙΝΙΟΥ. Ε, σας ακούσουμε λοιπόν, είναι η ερώτηση, ας ακούσουμε λοιπόν την απάντηση της Κομισιόν. Είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές η ουσία είναι ότι οι βουλευτές από το Ρινιού υπέβαλαν μια ερώτηση τον Σεπτέμβριο, αλλά δεν είχαμε λάβει γραπτή απάντηση μέχρι στιγμής εντός ε, της ε, προθεσμίας των έξι εβδομάδων. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του κανονισμού, άρθρο 138 για την ακρίβεια. Αφού δεν υπάρχει λοιπόν γραπτή απάντηση, ε, ζητήθηκε από την Κομισιόν να μας δώσει τις πληροφορίες ε, προφορικά στην συνεδρίαση. Και δίνουμε άρα τον λόγο στον κύριο Μάρκ Σόλωνα, επικεφαλής ε, της σχετικής μονάδας της Κομισιόν Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και στην κυρία Κλέρχαουτ για να μας δώσουν τις σχετικές πληροφορίες και έτσι οι βουλευτές που έκαναν την ερώτηση θα μπορέσουν να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για να ακούσουν και οι υπόλοιποι βουλευτές αλλά αυτό έχει προγραμματιστεί σε 30 λεπτά από τώρα οπότε προτείνω ναι με συγχωρείτε έχει προγραμματιστεί για να διαρκέσει 30 λεπτά να περιοριστείτε σε ένα λογικό χρονικό διάστημα. Πρότεινω δύο λεπτά για τον κάθε βουλευτή. Ας ακούσουμε όμως πρώτα την Κομισιόν. requested by this written question by the LIBE members. The Commission. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. όσον αφορά την ε, καθυστέρηση στην απάντηση. Ζητούμε ειλικρινώς συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση σε αυτό το ευαίσθητο και σημαντικό θέμα. Σας διαβεβαιώ ότι η πρόεδρος Φοντερ Λάιν ζήτησε από όλους τους επιτρόπους ε, να την ιδιαίτερη προσοχή στις απαντήσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, έχει ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης της γραπτής απάντησης. Για την ερώτηση τώρα και την διαδικασία αξιολόγησης. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η Κομισιόν δεν είναι σε θέση να σχολιάσει ε, το περιεχόμενο μιας ε, έκθεσης ε, αξιολόγησης η οποία είναι περιορισμένη. Δεν μπορώ λοιπόν να επεκταθώ επί της ουσίας έκθεσης. Μπορώ να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για τα διαδικαστικά βήματα που έχουν γίνει. Όπως ξέρετε, η επίσκεψη αξιολόγησης Σέγγεν στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε χώρα τον Νοέμβριο 2017. Η Κομισιόν ενέκρινε τη σχετική έκθεση τον Μάιο του 2018 και την απέστειλε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στις 16 Μαΐου 2018 η Κομισιόν παρουσίασε τα βασικά αποτελέσματα της αξιολόγησης στην ομάδα εργασίας ε, εποπτείας Σέγγεν. Η ομάδα εργασίας Σέγγεν συζήτησε την έκθεση τον Ιούνιο του 2018 και συζήτησαν και δύο επιλογές. Η πρώτη ήταν δεδομένης της ε, σοβαρότητας ε, του πράγματος. Δεν μπορούσε υπάρξει επανόρθωση, άρα θα έπρεπε να αποσυνδεθεί το Ηνωμένο Βασίλειο από την βάση δεδομένων. Το δεύτερο ήταν να κάνει η Κομισιόν κάποιες συστάσεις και να δώσει την ευκαιρία στο Ηνωμένο Βασίλειο να προτείνει ένα σχέδιο δράση. Το Συμβούλιο αποφάσισε να μην αποσυνδέσει το Ηνωμένο Βασίλειο και ζήτησε από την Κομισιόν να συνεχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης δίνοντας την ευκαιρία στο Ηνωμένο Βασίλειο να προτείνει ένα σχέδιο για διορθωτικές δράσεις. Παρ' όλα αυτά, η Κομισιόν πάγωσε προσωρινά την διαδικασία αξιολόγησης το φθινόπωρο του 2018 δεδομένων των διαπραγματεύσεων του Brexit και των προετοιμασιών για ένα σενάριο αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Τώρα η Κομισιόν εξετάζει το αν θα συνεχίσει την διαδικασία αξιολόγησης καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο θα χρησιμοποιεί το σύστημα κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020 περίοδος που μπορεί να παραταθεί κατά ένα ή δύο έτη. Μάλιστα. Αυτή είναι η δήλωσή σας. Εντάξει. Τελειώσατε. Έχετε να πείτε κάτι άλλο. Όχι. Για την ώρα όχι. Ας ακούσουμε λοιπόν τους βουλευτές της ομάδας Ρίνιου. Προτείνω καθώς το ερώτημα υποβλήθηκε από 20 βουλευτές 15-16 ε, προτείνω η κυρία Ίνετφελντ να το παρουσιάσει. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία διόρθωση στην Κομισιόν αναφέρθηκε σε καθυστέρηση. Δεν είναι καθυστέρηση, δεν έχει απαντήσει. Ε, μου προξενεί έκπληξη η απάντηση της ε, Κομισιόν. Ε, πρώτα απ' όλα λέτε ότι δεν θέλετε να σχολιάσετε ένα εμπιστευτικό έγγραφο. Το έγγραφο έχει δημοσιευτεί. Και θα πρότεινα σε όλους τους συναδέλφους να το διαβάσουν. Είναι σοκαριστικό πραγματικά. Κάθε σελίδα αναφέρεται σε πολύ σοβαρές ελλείψεις στην εφαρμογή του συστήματος Και πρέπει να θυμόμαστε αγαπητοί φίλοι, να μην για μια χώρα η οποία δεν είναι μέλος της Σέγγεν γιατί δεν θέλει να είναι μέλο τη Σέγγεν, ούτε καν τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, από την καλή μα την καρδιά, του δώσαμε πρόσβαση. Και ε, κάνουν ό,τι θένε εκεί μέσα. Ε, δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώ. Δηλαδή, διάβασα την έκθεση και πάλι είναι. σοκαριστική. Και το ότι κάνουν παράνομα αντίγραφα. Δηλαδή, ε, έτσι κατέληξε στα μήμια και κάναμε τις ερωτήσεις. Σε κάθε σελίδα, το βλέπετε, υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις, όπως τα λέει η ομάδα αυτή. Ε, εγώ θα έλεγα ότι είναι εσκεμμένες παραβιάσεις και καταχρήσεις του δικαιώματος πρόσβασης στο σύστημα και μια ηρωνική παραβίαση μάλιστα είναι το ότι δεν υπάρχει αμοιβαιότητα. Δηλαδή εμείς δίνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόσβαση σε ένα σύστημα στο οποίο επισήμως δεν είναι μέλη, υποθέτοντας ότι θα συνεισφέρει στη δική μας την ασφάλεια γιατί θα συνεργαστούν μαζί μας σε ζητήματα καταπολέμησης τρομοκρατίας και μετά δεν το κάνουν. Δηλαδή, μας δώσατε εδώ δύο επιλογές. Είτε να αποσυνδέσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο, είτε να τους δώσουμε χρόνο να προτείνει ένα σχέδιο για διορθωτικές δράσεις διορθωτικές. Εγώ ξέρω ποια είναι η επιλογή μου. Αποσύνδεση. Σήμερα. Δηλαδή, αν κάποιο συμπεριφέρεται με τρόπο εγκληματικό, του βάζουμε φυλακή. Δεν λέμε θα σου δώσουμε λίγο χρόνο να κάνεις κάποιες διορθωτικές δράσεις. Όχι, παραβιάζει τον νόμο, πα φυλακή, τελεία. Ε, συνάδελφοι, πρέπει εδώ πέρα να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Γιατί, ε, ειλικρινά, έχει εδώ πέρα ε, το Κοινοβούλιο μια επιτροπή παρακολούθηση Σέγγεν. Εγώ δεν ήμουν ε, μέλος ποτέ. Ε, πώς δεν προέκυψε ποτέ αυτό. Δηλαδή, αν αυτά κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο και έτσι φέρεται η Κομισιόν, τι άλλες παραβιάσεις υπάρχουν στις άλλε χώρε. Σοκάρομαι πραγματικά. Συμπερασματικά λοιπόν. Η Κομισιόν δεν μας έχει ενημερώσει πλήρως. Αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες της ε, στο να διασφαλίσει την ακαιρεότητα και την ασφάλεια του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν. Αυτά τα διαβάζω μέσα από την έκθεση. Οπότε η Κομισιόν δεν ε, κάνει αυτό το οποίο έχει καθήκον απέναντι στους πολίτες. Δεύτερον, το Ηνωμένο Βασίλειο πώς θα το πούμε ευγενικά, δεν νοιάζεται για τις υποχρεώσεις του και όμως συνεχίζει να έχει πρόσβαση. Τρίτον, το κοινοβούλιο προφανώς επίσης δεν ασχολείται. Και τέταρτον, θα μπούμε προσεχώς σε διαπραγματεύσεις με το ΕΒ Βασίλειο για τη μελλοντική μας σχέση. Ε, δηλαδή, εάν έτσι βλέπει η Κομισιόν την τρέχουσα σχέση με το ΕΒ Βασίλειο όσο ένα ακόμα μέλος Δηλαδή, τι να πούμε για τη μελλοντική μας σχέση. Ε, για μένα Καμία πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Τελεία και παύλα. Και αν αυτή είναι η αξιοπιστία του εταίρου μας εδώ πέρα, πρέπει να είμαστε σαφείς. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους υπό αυτές τις συνθήκες. Ευχαριστώ κυρία Ιντφελτ. Η κυρία Ντάλη ζήτησε το λόγο. Thank you. Sorry, didn't... Ευχαριστώ και συγγνώμη, δεν περίμενα να δώσω το λόγο τόσο γρήγορα. Συμφωνώ απόλυτα με την ε, γραπτή ερώτηση. Και είμαι πολύ απογοητευμένη με την προφορική απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει σχετική έρευνα σε κάθε περίπτωση. Δεν έχουμε ακούσει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο όμως ως τώρα και αυτή η έρευνα θα πρέπει να περιλαμβάνει και έρευνα για το ποιος τα έδωσε την εντολή για τα δεδομένα αυτά, το κόστος, ποιοι ενημερώθηκα από την ε, κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, από ποιε εταιρείε ενημερώθηκαν και πραγματικά οι συνέπειε είναι πάρα πολύ σοβαρέ. Ε, αναφέρονται στις ε, σχόλια του πρώην Επιτρόπου Κέν και σε ό,τι αφορά τα πρακτικά βήματα τα οποία λήφθησαν για να αντιμετωπίσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο από αυτόν, αλλά και άλλα κράτη-μέλη, όπω είπατε, αντιμετωπίζουν προκλήσει εδώ. Αυτό είπατε. Ποια είναι αυτά τα κράτη-μέλη, θέλω να ξέρω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τα δηλώσει όλα αυτά για το πόσο τραγική είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ε, προστασία των βάσεων δεδομένων αυτών. Και το λέω αυτό ως μέλος της ε, Επιτροπής Παρακολούθησης του Σέγγεν. Είναι πραγματικά ειρωνικό το γεγονός ότι μιλάμε για μια τέτοια παραβίαση τέτοια και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δεν είχαν καν πρόσβαση, δεν είχαν μυριστεί το τι γινόταν. Ήταν πραγματικά ε, τραγική η έλλειψη των πληροφοριών σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Επίσης, σημειώνω ότι ο κύριος Κέιν είχε σχολιάσει το άρθρο αυτό και είχε πει ότι πρόκειται για απόρριτα στοιχεία τα οποία έχουμε για τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Όχι. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε απόρριτο επ' αυτόν. Το εσωτερικό α, έγγραφο έχει κυκλοφορήσει ευρέω. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη κοινοποίησή του. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ως απόρριτο και θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες αυτές. Ακριβώς γιατί ο κόσμος ο οποίος α, α, τελικά υπέστη παραβίαση των δικαιωμάτων θα πρέπει να έχει δικαίωμα προσφυγής. Κάτι άλλο που με ανησυχεί. Για τις αρχές των ΙΠΑ που ανησυχούμε ότι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά χρησιμοποιώντας το Patriot Act και άλλα δημοσχέδια. Αναφέρθηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και το Υπουργείο Εσωτερικών, τα αναφέρει όλα αυτά γιατί εκεί τίθεται θέμα ιστορικών διεργασιών και πνευματικών δικαιωμάτων. Αν εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει να σχολιάσει τίποτα, είναι εξοργιστικό. Δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία για κλεμμένε βάσει δεδομένων που περιλαμβάνουν ιδιωτικέ πληροφορίε για ιδιώτε σε μια χώρα η οποία σε σύντομα θα είναι τρίτη χώρα. Κυρία Ντάλη, ναι, ολοκληρώστε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πραγματικά θα πρέπει να ανέλθει στο ύψο των περιστάσεων. Θα θέλαμε να, να ξέρουμε λοιπόν κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βγει και έχει υποβάλει ένσταση για αυτό το θέμα των ε, πνευματικών δικαιωμάτων που ισχυρίζεται το Ηνωμένο Βασίλειο και κατά πόσον υπάρχουν αντίτυπα των κλεμμένων αυτών ε, δεδομένων και τι γίνεται για να, υπάρξει, να μην υπάρξει περαιτέρω διάδοση των πληροφοριών αυτών, των δεδομένων αυτών. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απάντηση. Ναι, Ευχαριστώ. Η κυρία Ζίπελ έχει το λόγο. Ζίπελ. Αλλά σας θέλουμε παρακαλώ μην υπερβαίνετε το χρόνο που δικαιούστε γιατί θα έχουμε πρόβλημα τα υπόλοιπα σημεία. Ευχαριστώ και να ξεκινήσω με μια γενική παρατήρηση. Γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα το οποίο καταδεικνύει με σαφήνεια ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να εστιάζονται μόνο Στι νέε νομοθεσίε. Όχι. Θα πρέπει να δαπανούμε πιο πολύ χρόνο στη σωστή υλοποίηση και εφαρμογή τη ήδη υφιστάμενη νομοθεσία. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο κενό. Είναι σαφέ. Τα δεύτερον, υπογραμμίζω όλα όσα είπε η συνάδελφο Σοφίντφελτ και θα ήθελα να επανέλθω σε δύο σημεία τα οποία ανέφερε. Να τα θέσω προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιε είναι οι γενικέ συνέπειε. Δεν αρκεί να λέμε ότι α, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά για κάποια άλλα κρατημέλη. Τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα, τι θα κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση, να διορθώσουμε την κατάσταση και να βεβαιωθούμε ότι όλα πλέον θα ε, εφαρμόζονται σωστά και να ζητήσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθει στο θέμα αυτό και να μας υποβάλει αναφορά στην Επιτροπή μας, δηλαδή για το ποιε είναι οι συνέπειες και ποια είναι τα ευρήματά τους, τα παρίσματά τους. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις μοναδικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θυμάμαι ότι πολλοί έλεγαν τι σημαντικό που είναι να έχουμε στενές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο για θέματα ασφάλειας. Τι σημαίνει όμως αυτό. Προφανώς τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται προ παράνομου σκοπού, με παράνομο τρόπο. Και να τα πάμε και λίγο πιο μακριά, αν θέλετε. Η πρόσβαση στην βάση δεδομένων του Σέγγεν ενδεχομένω να υποδεικνύει παρόμοια προβλήματα με άλλε βάσει δεδομένων. Αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν μιλάμε για τις μελλοντικέ μας σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπράιαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, η χρήση της βάσης ε, δεδομένου από το Ηνωμένο Βασίλειο ε, εν, μέρη είναι παράνομη, αλλά είναι και ανεπαρκής. Αυτό να το υπογραμμίσουμε, νομίζω. Δεν μιλάμε μόνο για τεράστια παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτική σφαίρα, αλλά και για θέματα ασφάλειας το Ηνωμένο Βασίλειο δεν κάνει συγχρονισμό και ενημέρωση τη βάση δεδομένων. Δηλαδή, αν γίνεται καταχώρηση κάποιων συλλήψεων, δεν θα φαίνονται στι ε, βάσει δεδομένων και μπορεί ένα υποπτό ε, κατηγορούμενο να διαφύγει μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου. Και αυτό είναι βασικό πρόβλημα. Ουσιαστικά χειραγωγούν τι καταχωρήσει αυτέ και δεν ε, κάνουν αυτά που ζητούν οι αστυνομικέ υπηρεσίε. Αυτό συνεπάγεται τεράστιους κινδύνους για την συλλογική μας ασφάλεια. Και άρα θέλω να υποδείξω το εξή. Καταρχάς, η καθυστέρηση για την, στην απάντηση της ερώτησης αυτής είναι παράδεκτη. Είναι παραβίαση των κοινοβουλευτικών κανόνων. Και κατά δεύτερον, η άρνηση να απαντήσουν σήμερα προφορικά και πάλι είναι κάτι το παράδεκτο. Ο κανονισμός προβλέπει με σαφήνεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται, υποχρεούται να απαντεί να απαντά σε ερωτήσεις αυτές. Αυτά τα έγγραφα δεν μπορούν να είναι απόρριτα γιατί έχουν να κάνουν με παραβίαση του κοινωτικού δικαίου και δεν μπορούν να τα στερούν από την ομάδα παρακολούθησης. Όπως είπε η Σόφι Ιντφέλτ, όντως θα πρέπει να αναστείλουμε, να σταματήσουμε την πρόσβαση του ε, στη βάση δεδομένων. Να μην συνεχίσει προφανώ το Ηνωμένο Βασίλειο να χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων υπό το νέο καθεστώ και να μα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν απαντήσετε και δεν απαντάτε στο πλαίσιο αυτό λόγω εμπιστευτικότητα. Μήπω μπορεί να γίνει μια ακρόαση και κλεισμένων των θυρών για να υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο να μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Ενημερώστε μας λοιπόν τι ακριβώς ε, χρειάζεστε, υπό ποιους όρους, για να υπάρξει ένας διάλογος, μια ανταλλαγή ε, επ' γιατί δεν πρόκειται να τη γλιτώσετε και να σας αφήσουμε να μην απαντήσετε καθόλου. Ωραία και για να ολοκληρώσουμε ε, τη συζήτηση θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Ιντφελτ και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Ιντφελτ πρώτα. Δεν έχω και πάρα πολλά να προσθέσω. Μία επιπρόσθετη ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσω, γιατί αυτές οι παραβιάσεις ήδη είχαν διαπιστωθεί το 2015 και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2017 διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε αντιμετώπιση των παραβιάσεων αυτών. Γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξεκίνησε άμεσα τη διαδικασία αποσύνδεση από το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί δεν είχαμε καν οποιαδήποτε πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά θέματα ασφάλεια. Για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέχισε να δίνει πρόσβαση στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον δεν ήταν πρόθυμοι και δεδεθμένοι να αντιμετωπίσουν τι παραβιάσει αυτέ. Δεν μιλάω για ανεπάρκειε, ήταν παραβιάσει, ήταν ηθελμένε. Γιατί λοιπόν συνέχισε να δίνει πρόσβαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα. Ε, ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλει να ξαναλάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά κάποιες εικασίες που έγιναν, κάποια συμπεράσματα που βγάλατε, θα ήθελα να τονίσω ότι ε, το άρθρο που αναφέρεται δεν ανταποκρίνεται στο το άρθρο του Observer δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της έκθεσης για τις επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων ΣΥΣ ε, και η συνεργασία με ιδιωτικέ εταιρείε σε οποιαδήποτε θέματα που αφορούν το ΣΥΣ εμπίπτουν στον κανονισμό για το ΣΥΣ και τη συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις του κανονισμού, κυρίως Εκείνε που αφορούν την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων. Επιπλέον, ο κανονισμό για το σύστημα πληροφοριών Schengen ε, προβλέπει ότι τα δεδομένα που έχουν τύχει επεξεργασία ε, ε, από τη βάση δεδομένων δεν μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Οπότε η διεθνει οργανισμους οποτε η κυβερνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να ζητήσει από, από τις επιχειρήσει, ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεδομένα που έχουν λάβει από το ΣΥΣ δυνάμει του νόμου Patriot των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως σας είπα, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε την έκθεση αυτή. και μία παραβίαση των κανόνων για, την, για τη μετάδοση πληροφοριών δεν οδηγεί άμεσα στην αποσύνδεση. Και το γεγονός ότι ένας δημοσιογράφος συνέταξε ένα άρθρο, δεν επηρεάζει ε, το, το καθεστώς της έκθεσης ε, ως ε, απόρριτου εγγράφου. Οπότε, ήδη το Μάιο του 2018 έγινε συζήτηση στην ομάδα ελέγχου του Σέγγεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει γίνει και σχετική συζήτηση με το Συμβούλιο. εκεί συζητήσαμε την έκθεση, γιατί εκεί ήταν η κατάλληλη ευκαιρία και το κατάλληλο φόρουμ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει τις εκθέσεις αξιολόγησης μετά την έγκρισή τους από τους αρμόδιους φορείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ολοκληρώσετε? Όχι. Και το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να σας επισημάνω και να σας υπενθυμίσω είναι ότι η χορήγηση πρόσβασης ε, στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν για το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ω εκ τούτου, δεν απόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει απόφαση για την αποσύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου από, την, ε, το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Ε, το, η ομάδα εργασία του Συμβουλίου επιλήφθηκε και οι δύο προτάσει που εξετάστηκαν στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου έγιναν από την ε, αρμόδια χώρα, από την ενδιαφερόμενη χώρα και όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Έχουμε πολλά θέματα. Οι συντονιστές θα μπορούσαν να εξετάσουν τη συνέχεια θα δώσουμε στο ζήτημα αυτό. Δεύτερον, η ομάδα ελέγχου ε, του Σέγγεν. Ε, θα αποφασίσουν οι συντονιστές πώς μπορεί να ενισχυθεί αυτή η συνέχεια και η έκθεση για το Σέγγεν θα μπορούσε να περιλαμβάνει και το σημείο αυτό. Η έκθεση της ΛΥΜΠΕ για το Σέγγεν. Και θα μπορούσαν οι συντάκτες της προφορικής ερώτησης να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους και να θέσουν το ζήτημα στους συντονιστές για να δούμε τι συνέχεια θα δώσουμε ώστε να ικανοποιηθεί καλύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προφορική μας ερώτηση. Αυτά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμετοχή και θα έλεγα να περάσουμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 7, την ε, αποστολή μας ε, στο Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας ε, στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, 30 με 31 Οκτωβρίου του 2019. Θα ακούσουμε την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης της αποστολής βάσει του ιστορικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιτρέπει σε κάθε επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθε δύο χρόνια να πραγματοποιήσει αποστολή τριμελή σε οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για του οποίου είμαστε αρμόδιοι. Η κυρία Κατερίνα Κινίτση ήταν η επικεφαλής της αντιπροσωπείας αυτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Κέντρο παρακολούθηση Ναρκωτικών και Τοξικομανία τη Λισαβόνα και θα μα παρουσιάσει το σχέδιο έκθεση τη αποστολή αυτή. Παρακαλώ κυρία Κινίτση, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. 30 και 31 Οκτωβρίου η Κομισιόν επισκέφθηκε στην Λισαβόνα το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ναρκωτικών και Τοξικομανίας ε, στην ε, πραγματικότητα λόγω διαφόρων προβλημάτων εκπροσώπησα εγώ το Κοινοβούλιο γιατί οι άλλοι συνάδελφοι της Επιτροπής ε, δεν μπόρεσαν να έρθουν. Άρα όλα αυτά, ε, ο διευθυντής εκεί πέρα, ο κύριος Αλέξης ε, Γκόσντελ μας παρουσίασε την εργασία τους με τρόπο εξαιρετικό και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και αυτόν και το προσωπικό του παρατηρητηρίου το οποίο μας παρουσίασε και ο, κύριος Φαβιο Περέιρα, επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερος και την ε, Γραμματεία και την κυρία Μόιρα Αντριανέλη, όπως επίσης ε, και τις συμβούλους των πολιτικών ομάδων οι οποίοι συμμετείχαν και πραγματικά συνεισέφεραν στην επιτυχία αυτής της αποστολής. Η αποστολή έγινε τρία χρόνια μετά από την προηγούμενη και στόχο είχε να δούμε τις εργασίες που γίνονται, την μεθοδολογία των εργασιών που είναι πολύ αποτελεσματική, αλλά και να δούμε την διάδοση του φαινομένου της τοξικομανίας και της χρήσης των ναρκωτικών στην Ευρώπη που περιλαμβάνουν και νέες ε, ουσίες ε, θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στο ότι την ε, πρώτη μέρα ασχοληθήκαμε με το θέμα της ε, εξάρτησης. Έχουμε λοιπόν μια αύξηση της χρήσης των ε, ναρκωτικών. ιδιαίτερα των οπιοειδών Βεβαίως η πιο διαδεδομένη ουσία παραμένει η κάναβη και η ηρωίνη δυστυχώς ε, είναι αυτή η οποία προκαλεί τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων, θάνατοι οι οποίοι από το 2017 ε, ανέρχονται σε 8.200 ε, που έφτασαν τους 9.400 εάν συνυπολογίσουμε Νορβηγία, και Τουρκία οι οποίε έχουν επίση μια συμφωνία ανταλλαγή πληροφοριών με το παρατηρητήριο. Η ιδιαίτερα ανησυχητική σκοπιά είναι η άνοδος των νέων αυτών ε, ουσιών, των συνθετικών όπιοειδών, ψυχοτρόπων ουσιών. Έχουμε λοιπόν έναν αριθμό και εκεί πέρα νεκρών, ο οποίο δυστυχώς αυξάνεται γιατί έχουμε νέε ε, ψυχοτρόπες ουσίες οι οποίες μπαίνουν στην αγορά, όπως το φεντανίλ, το οποίο είναι ένα αναλγητικό, ε, μια ουσία αναισθητική, η οποία κατά κανόνα χρησιμοποιείται στην ιατρική και στην κτηνιατρική, και η οποία όμως ε, δυστυχώς χρησιμοποιείται πλέον με τρόπο ακατάλληλο ως ναρκωτική, ως ε, ψυχοτρόπος ε, ουσία μέσω του παρανόμου εμπορίου στο διαδίκτυο γιατί και μια ελάχιστη δόση δυστυχώς ε, προκαλεί τεράστιες βλάβες και έχει πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο για την υγεία. Δυστυχώς όμως είναι πάρα πολύ εύκολη η εμπορία της γιατί όπως σας είπα είναι πολύ μικρές οι δόσεις. Έχουμε λοιπόν από το 2007 ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ε, το οποίο μέχρι στιγμής ε, έχει προβεί σε 1300 τέτοιες ε, ειδοποιήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε τις διαφορές ροές προέλευσης των ναρκωτικών ουσιών οι οποίες παραμένουν στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος. Οι χώρες είναι η Νότια Αφρική, η Βόρεια Αφρική, και Δυτική Ασία. Υπάρχουν όμως και νέες χώρες, η Ινδία και ιδιαίτερο η Κίνα, οι οποίες έχουν γίνει σημαντικές χώρες προέλευσης, παραγωγής δηλαδή, ε, σε επίπεδο μάλιστα βιομηχανικό σύμφωνα με το παρατηρητήριο ψυχοτρόπων ουσιών. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο πολύ χαρακτηριστικό το οποίο μας παρουσιάστηκε για το πώς ακριβώς χρησιμοποιούνται οι ναρκωτικές ουσίες στην Ευρωπαϊκή Επικράτη. Η δεύτερη μέρα αφιερώθηκε στην δραστηριότητα του ίδιου του παρατηρητηρίου σε θέματα προϋπολογισμού και οργάνωσής του έχει γίνει μια εξωτερική αξιολόγηση από την Κομισιόν η οποία προβλέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό κάθε έξι χρόνια είχε γίνει το 2007 και το 2018 και επιβεβαίωσε πως ε, λειτουργεί πάρα πολύ καλά το παρατηρητήριο και Επίσης ε, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όπως παραδείγματος χάρη βελτίωση της εικόνας του και της δουλειάς που κάνει προς τα έξω για να υπάρξει μεγαλύτερη διάδοση των πληροφοριών που αυτό παρέχει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σε σχέση με τα όσα γίνονται τώρα. Η εξωτερική αξιολόγηση δεν ε, μπήκε στο πώς ε, θα μπορούσε να επεκταθεί η δραστηριότητα του παρατηρητηρίου και σε άλλες εξαρτήσεις ε. όπως παραδείγματος χάρη αυτές που υπάρχουν από το αλκοόλ, τον τζόγο και το διαδίκτυο. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό για το 2020 αυτός παραμένει σταθερός και αυτό παρά το το κόστος του προσωπικού αυξήθηκε. Αυτό δεν έχει δημιουργήσει ε, δυσκολίες στη λειτουργία του καθώς έχει εξακολουθεί να παράγει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα δεδομένων των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων που έχει. Εν ολίγης, ε, κυρία Πρόεδρε, για να καταλήξω, μπορώ να σας πω πως ε, η Αποστόλη αφενός διαπίστωσε την ε, εξαιρετική λειτουργία του παρατηρητηρίου, ειδικά όσον αφορά την μεθοδολογία εργασίας που ακολουθεί και επαληθέψαμε, επαληθέψαμε πως Η εργασία αυτή στηρίζει τις ε, πολιτικές ε, στον τομέα των ε, ναρκωτικών ουσιών και στο εμπόριό τους δηλαδή παρέχει δεδομένα αξιόπιστα και συγκρίσιμα για το φαινόμενο των ναρκωτικών και της τοξικοεξάρτησης. Είναι λοιπόν σημαντικό να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός του και στο πλαίσιο των, διαπραγματεύσεων που γίνονται για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 2027 για να έχει επαρκή χρηματοδότηση και πιθανώς να αυξηθεί εάν αυξηθούν και οι αρμοδιότητες τους. Και θεωρούμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα της εργασίας του παρατηρητηρίου. Τέλος, ε, αυτό το οποίο είπα, βλέπουμε μια αύξηση δυστυχώς τα τελευταία χρόνια του φαινομένου της ε, τοξικοεξάρτησης ε, και όπως είπε και η Κατερίν Ντεμπόλ της Europol ακόμη μια φορά και αυτό το βλέπουμε και στην κοινή έκθεση του παρατηρητηρίου και της Europol που θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή μας τέλος Ιανουαρίου, το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών παραμένει μία από τις πιο επικερδείς δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος και τροφοδοτεί με τη σειρά του άλλες μορφές εγκλήματος. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε την πολιτική καταπολέμησης ε, των ναρκωτικών ε, που είναι πάρα πολύ σημαντική βέβαια στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας ε, καθώς αντιλαμβάνεσαι ότι αποτελεί μια απειλή για την δημόσια υγεία το φαινόμενο αυτό. Οπότε μπορώ να πω ότι ήταν μια αποστολή σημαντική η οποία ολοκληρώθηκε θετικά και ανέδειξε νομίζω την εξαιρετική δουλειά που γίνεται εκεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κινίτσι. Ευχαριστούμε θερμά για την διεξοδικότατη ενημέρωση που μας κάνατε και τον απολογισμό της αποστολής σας στην Λισαβόνα και χαίρομαι που το παρατηρητήριο λειτουργεί εξαιρετικά, με σωστή μεθοδολογία, με αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες και στοιχεία και φυσικά θα μπορούσε να βελτιωθεί με αύξηση του προϋπολογισμού. Και είναι σημαντικό ε, που μας είπατε ότι αυξήθηκε η τοξικομανία και χρήση ναρκωτικών και αυξήθηκαν δυστυχώς και οι θάνατοι από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Στα τέλη του Ιανουαρίου θα έχουμε και την έκθεση για αυτές τις ε, τρομερές και εγκληματικές πρακτικές που δημιουργούν τόσα προβλήματα ε, σε πάρα πολλές οικογένειες στις χώρες μας. Και αφορούν την υγεία και το μέλλον των ε, νέων που πέφτουν δυστυχώς σε πολλαπλές μορφές τοξικομανίας και τοξικοεξάρτησης. Αυτά. Θέλει κανείς το λόγο παρακαλώ. Υπάρχουν σχόλια. Όχι από ό,τι βλέπω. Ή μάλλον η συνάδελφος ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δα, διάβασα πρόσφατα την ε, έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, του παρατηρίου αυτού του 2018 για την αγορά ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πραγματικά είναι σοκαριστικό το έγγραφο, αλλά αποδεικνύει το εξαιρετικό έργο του παρατηρητηρίου. Βλέπουμε ότι η κοκαίνη έχει επανέλθει στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και η Πολωνία φαίνεται ότι είναι η μεγαλύτερη αγορά κοκαίνης στην Ανατολική Ευρώπη. Η έκθεση σημειώνει ότι οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να αναχαιτήσουν το φαινόμενο και έχουμε ρεκόρ κατασχέσεων. Η Πολωνία όμως μέχρι στιγμής έχει ε, καταγγείλει μόνο εννέα κατασχέσεις ε, για το 2017 και για τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε καν στοιχεία ε, υποβάλει. Μπορείτε να το σχολιάσετε, έχετε περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για το σημείο αυτό. Τι κάνει το κέντρο σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες εφαρμογής, τους πόρους. Βλέπουμε αυτά τα στοιχεία που μας δίνει η έκθεση για την Πολωνία. Τι μέτρα λαμβάνει το παρατηρητήριο για τα θέματα αυτά. Μάλιστα. Ο κύριος Σερβανίτης επίσης ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Sorry, καλή χρονιά. Ήθελα να σας πω από την καρδιά μου. Ε, είμαι από τους ε, άτυχους. Μια βαριά ίωση δεν μου επέτρεψε να πάω σε αυτό το ταξίδι και έχω όμως μια εμπειρία που θέλω να τη μοιραστούμε. Σε ό,τι αφορά στο κέντρο παρακολούθησης ναρκωτικών, καθώς 35 χρόνια, το είχα ξαναπεί πάλι σε αυτή την Επιτροπή, ασχολούμαι με το θέμα των εξαρτήσεων ως Αντιπρόεδρος του Δημόσιου Φορέα Θεραπευτικών Κοινοτήτων στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σας πω ότι το κέντρο είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τα θεραπευτικά προγράμματα ε, μεικτά προγράμματα, στεγνά προγράμματα, τα θεραπευτικά προγράμματα των χωρών μας και οι δομές αυτές αξιοποιούν όλη αυτή τη γνώση για να χτίσουν εθνικές στρατηγικές σε ό,τι αφορά στο θέμα των εξαρτήσεων και βεβαίως των ναρκωτικών ουσιών. Γνωρίζω και προσωπικά τον ε, Αλέξη, τον διευθυντή δηλαδή, γνωρίζω προσωπικά και το προσωπικό πάρα πολλού, τους εμπιστεύομαι απόλυτα. Θέλω να σας πω ακόμα δύο πράγματα που μπορεί να βοηθήσουν γενικότερα τη δουλειά μας αυτή την πενταετία εδώ. Σε αυτό που είπε πριν από ένα λεπτό η συνάδελφο, τι κάνει το κέντρο, πρέπει να σημειώσω και ένα άλλο ζήτημα στι εξαρτήσει. Έχουμε ένα νέο φαινόμενο στην ε, Ευρώπη και ιδιαίτερα σε χώρε που βρίσκονται σε οικονομική κρίση, την πολυτοξικομανία. Δηλαδή, φτωχά στρώματα του πληθυσμού, ενώ πριν από ένα διάστημα είχαν ε, χρήση μια ουσία, χρησιμοποιούν αλκοόλ, αμφεταμίνες, ε, ηρωίνη, κοκαίνη, ό,τι βρουν στην αγορά. Αυτό δημιουργεί μια νέα κατάσταση στον κόσμο των χρηστών όπου δημιουργούν και σοβαρά προβλήματα ψυχολογικών και ψυχιατρικών προβλημάτων. Έχουμε μια νέα, ε, θα έλεγα, τάξη χρηστών στην ίδια βεβαρημένη προβληματική ομάδα χρηστών. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι... Α, βεβαίως έχουμε πολλά ένταση πια και στη δική μου χώρα στην Ελλάδα συνθετικών ναρκωτικών και βεβαίως θεωρώ, το έχω προτείνει και στους ανθρώπους του κέντρου, ότι πρέπει να ανοίξει λίγο το κέντρο παρακολούθησης, να είναι εξαρτήσεων, διότι ε, κλειδώνει το ένα πάνω στο άλλο η εξάρτηση του τζόγου με την εξάρτηση από ουσίες του αλκοόλ και έχει άμεση σχέση και αυτό που είπα με την πολιτικοσκομανία. Θα έλεγα τέλος ότι πολλές φορές αυτά τα πολύ καλά εργαλεία που έχει η Ένωση όπω είναι το Κέντρο Παρακολούθηση Ναρκωτικών. Εμεί είχαμε προτείνει και αύξηση των κονδυλίων για την παροχή υπηρεσιών προ εμά από το κέντρο. Πρέπει να κατευθύνουμε και την πολιτική μα και σε ενιαίο, σε ένα βαθμό γραμμή για το πώ βλέπουμε εμεί τι εξαρτήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να υπάρχει αυτό που λέμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ε, μοντέλο για το πώ θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Σα λέω ότι και στη δική μου χώρα, φαντάζομαι και στι δικέ. Ναι, ναι, ένα λεπτό μου ο Χρήστης πια, Πρόεδρε, είναι από τα 12 του χρόνια. Και αυτό είναι, είναι φοβερό. Thank you. Σας ευχαριστώ. Αν δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι θερμότατα την κυρία Κινίτσι για την ε, εξονυχιστική ενημέρωση που μας έκανε της αποστολής και ευχαριστώ και τον κύριο Ερβανίτη γιατί πραγματικά με την εμπειρογνωμοσύνη του έδειξε πολλά χρήσιμα ζητήματα. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, το σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης που αφορά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ad hoc αντιπροσωπείας της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που έγινε στη Μάλτα 2 και 3 Δεκεμβρίου 2019 ε, και της οποίας επικεφαλής ήταν η κυρία Ιντβέλτ που θα μας κάνει και έναν απολογισμό της αποστολής αυτής. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και το έργο σας στη Μάλτα εκ των προτέρων πριν καν ακούσω την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ και θα είμαι μάλλον σύντομη να σας δώσω μία σύντομη επισκόπηση του τι έκανε η αντιπροσωπεία. γιατί από την επίσκεψη του Κοινοβουλίου ε, έχει συζήτηση το Κοινοβούλιο και υπάρχει ένα ψήφισμα από το Δεκέμβριο, το 18 Δεκεμβρίου. Έχει περάσει λοιπόν καιρός, αλλά παρόλα αυτά καλό είναι να ενημερώσουμε τα μέλη της Επιτροπής πώς προέκυψε αυτή η προσωπία, αυτή η επίσκεψη και τι έκανε ακριβώς. Να ευχαριστήσω καταρχάς τη Γραμματεία γιατί πραγματικά εργάστηκαν σκληρά, έκαναν θαύματα για να διοργανώσουν αυτή την επίσκεψη, γιατί μέσα σε ημέρες κατάφεραν να τα οργανώσουν όλα και μάλιστα ήταν και πολύ καλό το πρόγραμμα και πραγματικά σας ευχαριστώ. Ο λόγος για τον οποίο ε, επισκεφτήκαμε τόσο άμεσα τη Μάλτα ήταν ότι υπήρξαν ε, δραματικές εξελίξεις ε, αναπάντεχες σε ό,τι αφορά την αστυνομική έρευνα για την δολοφονία της Δάφνη Καρουάνα Καλίτσια Είχαμε ήδη προγραμματίσει επίσκεψη στη Μάλτα, αλλά αργότερα προγραμματιζόταν αρχικά. Αποφασίσαμε όμω να είμαστε παρόντε στην παρούσα, στην φάση εκείνη, για δύο λόγου. Καταρχά, για να ενημερωθούμε από πρώτο χέρι σχετικά με τα τεκτενόμενα και θεωρώ ότι μια τέτοια επίσκεψη δεν έχει σκοπό μόνο να συλλέξει πληροφορίε και να μιλήσει με τον κόσμο, αλλά για να στείλουμε και ένα σαφέ μήνυμα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μα νοιάζει, ότι ανησυχούμε και ότι είμαστε παρόντες και ότι παρακολουθούμε. Είχαμε συναντήσεις λοιπόν με τον ε, Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Δικαιοσύνη, τον... την Τρίτη το πρωί, με τον Πρόεδρο επίσης, με τον Γενικό Εισαγγελέα, με τον υπεύθυνο της αστυνομική ε, δύναμης, ε, με την ομάδα του που διερευνά τη δολοφονία συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, με τον πρόεδρο της Αντιπολίτευσης, με τον διαμεσολαβητή. Είχαμε συνομιλίες με εκπρόσωπους της οικογένειας της ε, κυρίας Καρουάνα Γκαλίτσια, με ακτιβιστές, δημοσιογράφους, ΜΚΟ και με το επιμελητήριο των ε, δικηγόρων και ήταν πραγματικά υπερπίδες το πρόγραμμα και μας έδωσε μια πολύ ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης. Σε ό,τι αφορά τα πορίσματά μας τώρα, ένα βασικό πόρισμα, το προφανές, ότι επιτέλους υπήρχε σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά την έρευνα για την τηλεφωνία αυτή, αλλά και ανησυχητικό το γεγονός ότι υπήρχε έλλειψη πρόοδου σε ό,τι αφορά την ε, διερεύνηση ατόμων που προφανώς ήταν άτομα ευαίσθητα. Έγινε λοιπόν κάποια πρόοδος από την επίσκεψή μας και μετά, αλλά διαπιστώσαμε ότι υπήρχε έλλειψη ε, πρόοδου σε σημαντικά ζητήματα. Ανησυχούμε επίσης και το είπαμε αυτό σε ό,τι αφορά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ανακοίνωσε την παρατησή του, προβλέπεται σε λίγες ημέρες, αλλά είχαμε την αίσθηση γενικά, και εγώ έχω την έντονη προσωπική αίσθηση, ότι έμεινε στη θέση του για κάποιες εβδομάδες και αυτό πραγματικά απειλούσε ιδιαίτερο στην ακυριότητα των ερευνών και κυρίως ότι όσα μας είπε δεν μας ικανοποίησαν. Καλώς ορίσαμε επίσης την ε, διεθνή ανεξάρτητη έρευνα η οποία έχει ξεκινήσει από τότε και έχει οδηγήσει σε νέες μαρτυρίες, σε νέα αποδεκτικά στοιχεία. Σημειώσαμε επίσης τον πολύ θετικό ρόλο και την παρουσία της Europol. Σημειώσαμε επίσης ότι μετά τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας ε, ξεκίνησε να τηρούνται αυτά που ανέφερε. Χαιρόμαστε γι' αυτό που ξεκίνησε τουλάχιστον αυτή τη δικασία. όπως σας είπα, το γεγονός ότι δεν υπήρχε πρόοδος στις έρευνες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος κτλ. Μας ανησυχεί. Μας ανησυχεί επίσης το γεγονός ότι δεν υπάρχει ελευθερία στα μέσα ενημέρωση και η ασφάλεια των δημοσιογράφων δεν είναι κάτι το οποίο εξασφαλίζεται. Προφανώς αυτά πάνε χέρι-χέρι. Και τέλος, βάσει των πορισμάτων της αποστολής και των πορισμάτων των προηγούμενων αποστολών, και προηγούμενων διαδικασιών παρακολούθησης. Το ψήφισμα το οποίο εγκρίναμε, επαναλάβαμε, όπως επαναλάβαμε και εκεί επί τόπου, την έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο κατευθείαν με την ε, κυβέρνηση της Μάλτας για το νομοθετικό πλαίσιο. Και ξέρω ότι αυτό ακόμα δεν έχει γίνει, παρά το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει ανησυχίες, έχει αποστείλει γραπτή επιστολή στη Μαλταζική κυβέρνηση αυτό φυσικά είναι ακόμα καλύτερο από αυτά που είχε κάνει η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δυόμιση χρόνια. Άρα κάτι κινείται στην όλη υπόθεση, αλλά όλα αυτά είναι πολύ διστακτικά. Και τέλος, μετά την επιστροφή μας Γράψαμε δύο επιστολές. μία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το μήνυμα αυτό ακριβώς και προς το Συμβούλιο, γιατί μετά από κάποιε ημέρε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συναντήθηκαν στα πλαίσια συνόδου. Και μιας και ένας από αυτούς ήταν ο κύριος Γιώζεφ ε, Μουσκάτα, καλέσαμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσει τα θέματα αυτά και νομίζω ότι ε, δεν όντως μας αγνόησε το Συμβούλιο ως ήθιστε. Δεν είχαν καν την ε, τυπική ευγένεια να στείλουν μια απάντηση στην επιστολή μας για να ενημερωθούμε τουλάχιστον για τους λόγους για τους οποίους αρνήθηκαν να θέσουν το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω. Να ευχαριστήσω τα μέλη τη αντιπροσωπεία, γιατί καταρχά. ήταν πολύ γρήγορα διαθέσιμη τελευταία στιγμή πραγματικά και πιστεύω ότι παρά το γεγονό ότι είμαστε από διαφορετικό πολιτικό υπόβαθρο ο καθένας μας και έχουμε διαφορετικές πολιτικές ευαισθησίες, τελικά συνεργαστήκαμε σε πνεύμα συναδελφικότητας και επικοδομητικής συνεργασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι λοιπόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ιντφελτ για την παρουσίαση. Κυρία Ιντφελτ, όπως είπατε, όπως φάγατε, αναγκάστηκα να φύγω από το Προεδρείο γιατί είχα άλλη μια ανηλυμένη υποχρέωση. Ευχαριστώ λοιπόν την συνάδελφο, την αντιπρόεδρο, την κυρία Πάγασα Σαουρτουντούα για το γεγονό ότι με αντικατέστησε. Και φυσικά να εκφράσω κι εγώ την εκτίμησή μου για τη δουλειά που έκανε η γραμματεία. Πραγματικά. Για να προετοιμάσει, να διοργανώσει την επίσκεψη αυτή. Αυτή η επίσκεψη τελευταία στιγμή στη Μάλτα της Επιτροπής μας ε, μπόρεσε να λάβει χώρα και να κάνει και τη δουλειά της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για όλη αυτή τη διοργάνωση. Τελευταία στιγμή πραγματικά. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο έργο. Υπήρξε μεγάλη πίεση. Τώρα, να ακούσουμε και τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας. Όσοι είναι εδώ στην αίθουσα, Να ακούσουμε την κυρία Μέτσολα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τη Σοφή, να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας για την πολύ ειλικρινή συνεργασία. Και εμεί, ε, Σοφή, συμφωνούμε και εμεί ευχαριστούμε όλα τα μέλη της Γραμματείας που νυχθημερών ε, εργάστηκαν για να διοργανώσουν την ε, αποστολή αυτή, η οποία ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη. Από την αποστολή λοιπόν αυτή και μετά από αυτά που είδαμε έκτοτε ήταν πραγματικά παράλογα. Πέρα από κάθε λογική και φαντασία ε, σε ό,τι αφορά την προσπάθεια να συγκαλυφθούν τα της δολοφονίας της Ντάφνη Καρβανεγκαλίτσια και πλέον να βρισκόμαστε σε χαρτογράφητα είδατα. Ο Πρωθυπουργό ανακοίνωσε ότι πρόκειται να παρατηθεί αυτή την εβδομάδα, αλλά τις τελευταίες 40 ημέρες όπως και τα τελευταία χρόνια. Προφανώς ε, αποδυνάμωσε τα θεσμικά μας όργανα και προσπάθησε να ξεγλιστρήσει. Ο κόσμος από την κοινωνία των πολιτών έχει εξηγηθεί στους δρόμους, ζητά λογοδοσία. Αυτό πραγματικά είναι το λιγότερο. Ο γιος της ε, Ντάφνης Καρουάνα Γκαλίτσια, ο Μάθιου, δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη χωρί αλλαγή. Είχε δίκιο. Και να σα πω ότι η αποχώρηση και η παρέτηση του Μούσκατ δεν πρόκειται να επιλύσει όλα τα προβλήματα τα οποία διαπιστώσαμε στην αποστολή. Έκτοτε λοιπόν ε, εγκρίναμε ένα ψήφισμα στην τελευταία ολομέλεια του Κοινοβουλίου που εντοπίζει διάφορα θέματα τα οποία θα πρέπει να επιλύσει η Μάλτα από τα νομικά κενά στο Σύνταγμά μας, από τον τρόπο που ορίζουμε ε, τα θεσμικά μας όργανα και διορίζουμε τους αξιωματούχους μας ε, και στο Κοινοβούλιο και τον τρόπο που καλύπτουμε τα προβλήματα στην αστυνομία μας, το θέμα των ε, διαβατηρίων που δίνει η Μάλτα σε άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη Μάλτα ή με την Ένωση. Προφανώς το Κοινοβούλιο θέλει να υποστηρίξει τον λαό της Μάλτας. Όταν θα ξεκινήσει, ελπίζουμε, ε, όταν θα ξεκινήσει την ανάκαμψή του από το καθεστώς του Μουσκάτ. Αλλά το θέμα σε τελική ανάλυση δεν είναι μόνο η Μάλτα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή τη, η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προάσπιση των δικαιωμάτων των λαών της Ευρώπης θα πρέπει να βελτιωθούν μέσω ενό νέου μηχανισμού κράτου δικαίου, μέσω ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να σταματήσουν τέτοια θέματα και να προστατευτούν οι δημοσιογράφοι. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι θα γίνει μια δραστική και γρήγορη αλλαγή. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσοι ε, βοήθησαν στην διενέργεια τη αποστολή αυτή Να ευχαριστήσω τους συναδέλφου που άνοιξαν τα μάτια τους και ήταν τι έγινε στη Μάλτα, τι γίνεται στη Μάλτα για την ευρεία υποστήριξη του ψηφίσματο αυτού τον προηγούμενο Δεκέμβριο σε ό,τι αφορά τη Μάλτα. Μας έστειλε αυτό ένα πολύ πολύ ηχηρό μήνυμα για αισιοδοξία και αλληλεγγύη προ το λαό τη Μάλτα. Δεν είμαι πεσημετιστρία. Ξέρω τι προβλήματα αντιμετωπίζει η χώρα μα, αλλά είμαι αισιόδοξη ότι θα ξεπεράσουμε. Ευχαριστούμε την κυρία Μέτσολα. Και τώρα να ακούσουμε τα άλλα μέλη τη αποστολή. Η κυρία Σίπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Όντως ε, πολύ άρον-άρον έγινε η οργάνωση και χάρη στο έργο της γραμματείας, το, το συμβούλων του προσωπικού ε, έγινε πολύ καλή προετοιμασία. Και μάλιστα ήδη την Παρασκευή μετά την αποστολή συντάχθηκε και το προσχέδιο της έκθεσης και πάλι χάρη στη συμμετοχή όλων αυτών των συναδέλφων και της γραμματείας και των ε, βοηθών μας. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω θερμά όλου του συναδέλφου που έλαβαν μέρο στην αποστολή, γιατί μπορεί να έχουμε πολιτικέ διαφορέ στο ΑΒ θέμα, αλλά το κλίμα μεταξύ μα ήταν μια χαρά, ήταν ε, πολύ θετικό και καταφέραμε να διεξαγάγουμε την αποστολή σε πολύ καλή ατμόσφαιρα και κλίμα. Ε, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση, τονίζω αυτά που είπε η Σόφιν Βέλτ. Δεν έχει νόημα να επισέλθουμε και πάλι σε λεπτομέρειες, γιατί παρόλο που εξετάζουμε ε, μόνο σήμερα την ε, έκθεση της αποστολής. Οι συνέπειες των αποτελεσμάτων αυτής της ε, έκθεσης ήδη συμπεριλήθησαν στα, στην έκθεσή μας του περασμένου Δεκεμβρίου, στο σχετικό ψήφισμα για τη Μάρτα. Και θα πρέπει βέβαια να εξασφαλίσουμε μια συνέχεια και να παρακολουθήσουμε τι συνέχεια έχει δοθεί. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία μεταρρύθμισης της νομοθεσίας και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει την πορεία των εργασιών αυτών για να διαπιστώσει πρόοδο. Επίσης, ε, στηρίζουμε τις έρευνες των ε, ε, διεκτικών αρχών. Ε, ιδιαίτερα κάποια διασυνοριακά ζητήματα που είναι απαραίτητα να διαθετηθούν για να σημειωθεί πρόοδο στην έρευνα. Σήμερα δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο γιατί ήδη λάβαμε μέρο στη συζήτηση που έγινε το Δεκέμβριο για τη Μάλτα, αλλά σίγουρα σε λίγου μήνε θα πρέπει να επανέλθουμε στα θέματα αυτά, όταν θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για τι μεταρρυθμίσει που έχουν ξεκινήσει και που ζητήσαμε να γίνουν. Ευχαριστώ θερμά όλου όσοι συνέβαλαν για να καταστεί δυνατή διεξαγωγή τη αποστολή και να στεφθεί με επιτυχία. Και θα πρέπει να δούμε τι διδάγματα θα αντλήσουμε από ό,τι μάθαμε και από τι αλλαγέ χρειάζονται. Και θα πρέπει να δούμε πώς ε, ε, λαμβάνεται υπόψη και η πολυφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελευθερία της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και θέματα διαφθοράς και εξεπλήματος χρήματος. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και αλλού δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς φυσικά να ξεχνούμε την ε, ιδιαίτερη κατάσταση της Μάλτας. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι η κατάσταση αυτή ξεπερνά τη Μάλτα. Κυρία Κάνκο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη γραμματεία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για την ανεκτήμητη συμβολή της στην επιτυχία της αποστολής και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία και την επικεφαλή στην κυρία Ίντβαλτ. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμότατα για την πολύ αγαστή συνεργασία που είχαμε και τον υψηλό επαγγελματισμό που ε, επιδείξατε σε αυτή την εξεταστική επιτροπή, στην εξεταστική μάλλον ε, αποστολή. Ε, διαπιστώσαμε πόσο σοβαρή και επίγουσα ήταν η κατάσταση και είναι, εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στη Μάλτα, όπως ε, τόνισε και η συνάδελφος Μετσόλα. Στόχος της αποστολής ήταν να συγκεντρώσει πραγματικά περιστατικά στοιχεία και ε, να τηρηθούν υψηλέ προδιαγραφές ε, της έρευνας ε, σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να παταχθεί η διαφθορά και το κράτο δικαίου να εφαρμόσει και στη Μάλτα και παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζω ότι η αποστολή και η ακόλουθη έκθεση να δώσει χρήσιμε πληροφορίε και στην ΛΥΜΠΕ, αλλά και στα άλλα θεσμικά όργανα. Σίγουρα η αποστολή αυτή δεν θα είναι το τέλο του έργου μα για την κατάσταση αυτή. Θα πρέπει να περάσει πολλής χρόνος για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του λαού προς τους θεσμούς ε, της Μάλτας. Πάντως, είναι σημαντικό τέτοιες αποστολές ε, να περιορίζονται στην ε, συγκέντρωση στοιχείων. Δεν είμαστε δικαστές. Είμαστε πολιτικοί και καθήκον μας στις αποστολές αυτές δεν είναι να διατρανώσουμε τις πολιτικές μας απόψεις, αλλά να συγκεντρώσουμε πραγματικά περιστατικά στοιχεία και φυσικά να απαιτήσουμε εφαρμογή του κράτους δικαίου. Και φυσικά χρειάζονται απαραίτητες διαδικασίες και στο μέλλον, ώστε να υλοποιηθεί το απολύτως απαραίτητο που είναι η εξασφάλιση τη δικαιοσύνη, η απονομή δικαιοσύνη για την οικογένεια της Δάφνης Καρουάνα που έχουν υποφέρει τα πάνδυνα πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε και νομίζω ότι η απόδοση δικαιοσύνη είναι αυτό που χρειάζεται. Βλέπω και τον κύριο Αρβανίτη από την ΚΟΕ στην αίθουσα. Παρακαλώ. Στην ΚΟΕ επιλέξαμε να έρθει στην αποστολή ο Στέλιος Κουλογλού διότι είχε ασχοληθεί δημοσιογραφικά ο ίδιος προσωπικά και εγώ δημοσιογράφος είμαι, είχα ασχοληθεί με άλλα θέματα και πιστέψαμε και η ΚΟΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ την αντιπροσωπεία να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ακόμα πιο πολύ το θέμα. Ε, μιλήσαμε με το Στέλιο, είναι σε επιτροπή για το Ιράν, γι' αυτό ε, θα σα πω δύο λόγια που συμφωνήσαμε να μεταφέρω στην Επιτροπή. Καταρχήν, θέλω και προσωπικά και ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει την ε, Σόφη, την επικεφαλή, διότι βοηθάει πάρα πολύ με τη σύνθεση και με τη λογική τη να δουλέψει πάρα πολύ καλή αυτή η ομάδα. Είμαστε πολύ ευτυχεί που δουλεύουμε μαζί τη. Και είμαι γκουε, είμαι άλλη πολιτική ομάδα. Θέλω να σα πω ότι η δολοφονία τη ε, Γκαλίσια μαζί με την δολοφονία του Σλοβάκου δημοσιογράφου Γιάν Κούσιακ νομίζουμε ότι πλήττει τον πυρήνα τη Ένωση. Μετά από χρόνια λοιπόν δημοσιογράφοι στην Ένωση δολοφονούνται για τι έρευνε ή εκβιάζονται ή πιέζονται μέσα από τις λογικές της διαφθοράς ή τα κανάλια της διαφθοράς στην πολιτική και την οικονομία μέσα στην Ένωσή μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξεχνιαστούν αυτές οι υποθέσεις. Η ιστορία της Μάλτας είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ε, με καλύπτει πλήρω η Σόφη για το πώ παρουσίασε τα πράγματα και οι άλλοι συνάδελφοι και νομίζω ότι αυτή η ιστορία τη Μάλτα θα είναι αρχή να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Thank you. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα, θέλει άλλος κανείς το λόγο? Όχι. Παρακαλώ, κυρία Σπούρεκ. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω πιο γενικά. Ε, πριν να ε, γίνω ευρωβουλευτή, ήμουν ε, αναπληρώτηρη επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Πολωνία. Ο καθηγητής Άνταμ Μπόλναρ, ο επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Πολωνία, χρησιμοποιώντα τις εξουσίε που του δίνει το Σύνταγμα, είχε τακτικές αντιδράσεις σε περίπτωση παραβίαση δικαίου στην Πολωνία. Και οι ευρωπαϊκές λύσεις ε, στην συγκεκριμένη περίπτωση κατέστησαν αναποτελεσματικές, γιατί όλο και περισσότερες χώρες φαίνεται ότι παραβιάζουν το κράτος δικαίου, μεταξύ αυτών και η Μάλτα. Θα πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε. Τι άλλο όμως μπορούμε να κάνουμε, ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα, αν το άρθρο 7, όπως έχουν δείξει τα παράδειγματα της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, δεν λειτουργούν. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει η νέα πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει τους υπέτειους στη δικαιοσύνη και πάνω απ' όλα να εφαρμοστούν μηχανισμοί και οικονομικοί για να αποτρέψουν άλλες χώρες από τέτοιες δράσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Η κυρία Ίντφελτ τώρα, πολύ σύντομα, γιατί συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Δεν, μπορεί, δεν μπορείτε να πει, ε, μιλάτε μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποιες περιπτώσεις. Το πρόβλημα είναι το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του για το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αρνείται να το κάνει. Και θα ήθελα ίσως να επαναλάβω ή να βάλω ένα αίτημα στον Πρόεδρο να υπενθυμίσει στο Συμβούλιο ότι είχαμε στείλει επιστολή τον Δεκέμβριο και ρωτήσαμε πότε θα λάβουμε απάντηση ε, γιατί δεν τέθηκε το ζήτημα της Μάλτας στη Σύνοδο Κορυφής. Μάλιστα, το μήνυμα ελήφθη. Θα ήθελα να σας πω ότι προτίθεμαι να είμαι παρόν στο πρώτο Συμβουλίο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που θα οργανώσει η Κροατική Προεδρία τον Ιανουάριο. Και νομίζω θα είναι ευκαιρία εκεί να υποβάλουμε αυτό το σημείο, δηλαδή πόσο σημαντικά είναι τα θέματα του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Μάλιστα, έχουμε και πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αίθουσα. Δεν ξέρω αν κάποιος από τη Γενική Διευθύνση Δικαιοσύνης θα ήθελε να προσθέσει κάτι για το σημείο αυτό ή όχι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καβριλιάδης από την Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι ο Ντιτιέ Ρέντερς έστειλε επιστολή στο Μαλτέζο Υπουργό Δικαιοσύνης επισημένοντα τα βασικά θέματα, το ανέφερε και η κυρία Ιντβελτ και φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγης την υπόθεση της Μάρτας ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όπως έχει κάνει μέχρι τώρα άλλωστε, και αν παραστεί ανάγκη θα λάβουμε και κατάλληλα μέτρα. Μάλιστα. Οπότε, ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό. Και δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Αυτά προς το παρόν. Ακούσαμε την παρουσία της έκθεσης ad hoc αντιπροσωπείας που έγινε στη Μάλτα και θα επαναλάβουμε την ευγνωμοσύνη μας προς όλες τις υπηρεσίες, βοηθούς, συμβούλους, γραμματεία που έβαλαν τα δυνατά τους για να σταθεί με επιτυχία αυτή η αποστολή. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η τρίτη ετήσια πανεξέταση της ε, ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ακούσαμε ε, τις παρουσίαση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον άλλο αρμόδιο φορέα, αλλά για τις 11 έχει προγραμματιστεί αυτή η παρουσίαση, σε 25 λεπτά από τώρα δηλαδή. Γι' αυτό προτείνω ένα σύντομο διάλειμμα και να συνεχίσουμε στις 11, αν δεν έχετε αντίρρηση. Εντάξει. Ραντεβού στις 11 λοιπόν και πάλι. 11 ακριβώς θα συνεχίσουμε. So, welcome back. Οπότε, καλώς ήρθατε και πάλι και σας ευχαριστώ. Και για όσους δεν ήταν εδώ σε 9, καλή χρονιά και πάλι. Και τώρα συνεχίζεται η συνεδρίαση. Περιμέναμε τους καλεσμένους μας, οι οποίοι ήρθαν για το σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης το οποίο αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας. την ετήσια έκθεση θα ακούσουμε λοιπόν την παρουσίαση της Κομισιόν και της, ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας ε, της Ιδιωτικής Ζωής. Θα ακούσουμε τον κύριο Μιχαήλ Φανφλέκερεν. Οκ. Α, ναι, ναι, μάλιστα. Τον Μπρούνο Καρέλη από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και από την Κομισιόν και την κυρία Λίζα Μαρή Λάγκε από το κρατήδιο της ΕΣΙΣ και τον κύριο Φρανσουά Πελερινή από την Γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. σας ακούσουμε πρώτα τον κύριο Τζεν Καρέλη από την Κομισιόν για την ετήσια έκθεση. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Καλή χρονιά σε όλους. Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα με τους ε, φίλους και συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων για να σας ενημερώσω για το πλαίσιο της προστασίας ε, δεδομένων και συγκεκριμένα τα όσα έγιναν ε, πέρσι 12 και 13 Δεκεμβρίου. Ξέρουμε ότι η ασπίδα αυτή καλύπτει τα εμπορικά δεδομένα που αφορούν τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, είναι κάτι το οποίο είναι πλέον αναπόφευκτο δεδομένων των διαφόρων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων από το εμπόριο μέχρι τις κοινωνικές συναναστροφές. Ακριβώς λόγω της μεγάλης ροής ε, δεδομένων δημιουργήθηκε αυτή η ασπίδα προστασίας τους. Ε, το πλαίσιο αυτό λοιπόν επεκτείνει την προστασία του γενικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν τα δεδομένα διασχίζουν τον Ατλαντικό. Αυτή τη στιγμή μέχρι, 5.000, ε, μέχρι αυτή τη στιγμή 5.000 εταιρείε έχουν δεσμευτεί να εφαρμόζουν αυτές τις διατάξεις και καθώς δεν υπάρχει σχετική ομοσπονδιακή νομοθεσία στη ΣΥΠΑ δεν θα υπήρχε προστασία χωρίς αυτήν την ασπίδα. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την συλλογή προσωπικών ε, δεδομένων από τις δημόσιες αρχές, μεταξύ των οποίων και τις αρχές εθνικής ασφαλείας. Έχουμε λοιπόν για πρώτη φορά ένα μηχανισμό σε διεθνές επίπεδο το οποίο έρευνα ε, καταγγελίες ε, άλλων δαπών, παραδείγματος χάρη Ευρωπαίων για τέτοια ζητήματα. Στο παρελθόν είτε δεν τους απασχολούσαν αυτά τα ζητήματα, είτε ήταν ζητήματα τα οποία συζητούνταν και κλεισμένων των θυρών και με μυστικότητα. Και βεβαίω αντιλαμβάνομαι πως έχετε σχετικέ ερωτήσεις, δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε, αλλά μην υποτιμούμε την ε, σημασία αυτών των υποσχέσεων. Μάλιστα η προστασία των δεδομένων έχει γίνει ένα σημαντικό κομμάτι του διαλόγου μας με τις ΙΠΑ και όσον αφορά και την προσβασία των δημοσίων αρχών. Παίζουν λοιπόν έναν σημαντικό ρόλο στον διάλογο αυτόν. Όπως ξέρετε, Είχαμε την, την εξέταση του θέματος ε, τον Οκτώβριο και μετά ακολούθησε η σύνταξη της έκθεσης. 14 Οκτωβρίου ήρθε ε, η Γενική Διευθύντρια, οπότε δεν θα τα επαναλάβω τα όσα είπε, αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι κάποιες σημαντικές πτυχές. Πρώτα απ' όλα να θυμόμαστε ότι όσον αφορά την συμμετοχή ε, μιλάμε για μια επιτυχία. Τα τελευταία χρόνια πάνω από 5.000 εταιρείε έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο αυτό και άρα δεσμεύονται από τις υποχρεώσει του. Ένας πολύ σημαντικό αριθμό. 5.000 εταιρείε είναι μεγαλύτερος αριθμός ε, από τις εταιρείε που είχαν ε, ενταχθεί στο προηγούμενο πλαίσιο σε 13 χρόνια. Αυτό περιλαμβάνει και αμερικανικές εταιρείες και θυγατρικές ευρωπαϊκών εταιριών στις ΗΠΑ. Ε, μιλάμε για εταιρείες ε, όπως η Aldi, η Randstad ή η Louis Vuitton. Επίσης είναι ένα βασικό κομμάτι ε, εργαλείο των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα στους εμπορικούς τους εταίρους ή στα υποκαταστήματα τους της ΕΠΑ. Έχουμε συγκεκριμένη πρόοδο σε σχέση με τις συστάσεις που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια και τις ανησυχίες που εξέφρασε το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων που είμαι σίγουρος ότι θα σας πει περισσότερα. Παραδείγματος χάρη έχει οριστεί επιτέλους μια μόνιμη διαμεσολαβητρία, αλλά η διαδικασία λειτουργεί και στην πράξη. Ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά πέρσι. Είχαμε την πρώτη καταγγελία, η οποία αντιμετωπίστηκε ικανοποιητικά επιπλέον επιβεβαιώθηκε το ότι η ίδια μεσολαβητρία δεν δρά μόνη της, αλλά σε συνεργασία με άλλες αρχές, όπως τις δικαστικές αρχές. Στην περίπτωση στην οποία είχε παραβιαστεί, παραδείγματο χάνει το άρθρο 702 του νόμου Φάιζα, που αφορά την παρακολούθηση δαπών στις ε, ΗΠΑ, το σχετικό δικαστήριο δίνει οδηγία στην αρμόδια υπηρεσία να διορθώσει την παραβίαση. Επίσης, ε, η Επιτροπή Παρακολούθησης των μυστικών υπηρεσιών ενημερώνεται συστηματικά και κάνει τις δικές της έρευνες. Έχετε την καλοσύνη να μιλάτε λίγο πιο σιγά γιατί ε, δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν οι διερμηνείς. Ναι, με συγχωρείτε. Επίσης, ε, ξεκαθαρίστηκε ότι ο Γενικός Επιθεωρητής των Μυστικών Υπηρεσιών ενημερώνεται σχετικά και κάνει ε, τις δικές του έρευνες, ο οποίος ενημέρωσε πράγματι και το Αμερικανικό Κογκρέσο για τις ε, καταγγελίες που οδήγησαν στην πρόσφατη παραπομπή του Αμερικανού Πρόεδρου. Επιπλέον, εάν μια τέτοια καταγγελία αποκαλύψει ότι τα δεδομένα αυτά έχουν συλλεχθεί παρανόμως θα διαγραφούν από τις αμερικανικές βάσεις δεδομένων και τα δεδομένα και οι αναφορές σε αυτά σε εκθέσεις. Οπότε θα μπορέσει να υπάρξει η διαγραφή των δεδομένων Ευρωπαίων πολιτών εάν έχουν συλλεχθεί παρανόμως από αμερικανικές υπηρεσίες. Θα αναφέρω αυτά γιατί ξέρω ότι αφορούν τις ερωτήσεις που έχετε κάνει στο παρελθόν και στα ψηφίσματά σας όσον αφορά τη λειτουργία του μηχανισμού. Επίσης, στην εξέταση είδαμε το πώς οι εταιρείε συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις αυτές και το πώς η συμμόρφωση αυτή ε, επιβλέπεται και επιβάλλεται. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε σημειώσει επίσης πρόοδο. Οι Αμερικανικές αρχές κάνουν περισσότερους προληπτικούς και συστηματικούς έλεγχους ε, Παραδείγματο χάρη το Υπουργείο Εμπορίου κάνει αιτησίους ε, ελέγχους ε, σε 30 εταιρείες οι οποίες αποτελούν μέλη της ασπίδας ε, προστασίας των προσωπικών δεδομένων και στην περίπτωση στην οποία δεν υπήρξε κάποια διορθωτική ενέργεια υπήρξαν ενέργειες από πλευράς Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου επιπλέον Καταλήξαμε στο ότι οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν περισσότερο τον μηχανισμό προσφυγής για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, το δικαίωμα παραδείγματος χάνει πρόσβασης ή το δικαίωμα διόρθωσης που είναι βασικά δικαιώματα με τους δικούς μας κανόνες. Οι πτυχές αυτές δεν αναφέρονται συχνά αλλά μιλάμε συχνά για την καθημερινή λειτουργία του πλαισίου και έχουμε λοιπόν απτά ωφέλη για τους Ευρωπαίους. Για να αξιολογήσουμε επίσης την αποτελεσματικότητα του πλαισίου πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η ασπίδα αυτή δεν λειτουργεί εν κενό, αλλά είναι μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου ενό μηχανισμού προστασίας δεδομένων στις ΕΠΑ και εκεί πέρα έχουμε δει θετικές εξελίξεις. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Υπάρχει σημαντική νομοθετική δραστηριότητα στις ΕΠΑ, κάτι το οποίο θα ξέρετε και ξέρετε αρκετοί από εσά που έχουμε συνεργαστεί σε τέτοια ζητήματα είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από λίγα χρόνια ότι θα συζητούσαν σοβαρά στο Κογκρέσο Ομοσπονδιακή τέτοια νομοθεσία. Η Καλιφόρνια πριν από λίγες μέρες ε, έθεσε ενισχύ Στη στιβάρους τέτοιου ε, κανόνες. Αυτά στο νομοθετικό επίπεδο, αλλά αυτό το οποίο είναι ακόμη σημαντικότερο είναι ότι η επιβολή αυτών των κανόνων έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια. Ας δώσω κάποια παραδείγματα. Έχουν επιβληθεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου πρόστιμα ε, μεταξύ των οποίων ένα πρόστιμο 5 δισεκατομμυρίων στο Facebook και 500 εκατομμυρίων σε μια άλλη εταιρεία και κατά τη Cambridge Analytica χάρη που απαιτήθηκε η διαγραφή όλων των δεδομένων των σχετικών. Ε, πρόκειται για πολύ σημαντική πρόοδο λοιπόν και ελπίζω σύντομα να δούμε σχετικά αποτελέσματα και σε αυτήν την όχθη του Ατλαντικού. Επίσης είχαμε ενδιαφέρουσες ε, περιπτώσεις ε, σε αυτόματες διαδικασίες, τους αλγόριθμους και συζητήματα που είναι πολύ σημαντικά για την τεχνητή νοημοσύνη, το η υπηρεσία για την στέγαση παραδείγματος χάριν ε, οδήγησε το Facebook στα δικαστήρια λόγω των στοχευμένων διαφημίσεων στον τομέα αυτών. Στον τομέα της εθνικής ασφάλειας επίσης ε, υπάρχει η, ε, λεγόμενη, υπάρχουν οι εκθέσεις του λεγόμενου P-Club του Συμβουλίου το οποίο εποπτεύει τα ζητήματα ιδιωτικής ζωής στις μυστικές υπηρεσίες ε, των ίπα, Κάτι το οποίο βεβαίως έχει απασχολεί συχνά και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στα ζητήματα εθνικής ασφαλείας έχουμε δει πως ο Γενικός Επιθεωρητής ε, και το Εποπτικό Συμβούλιο έχουν παίξει τον ρόλο τους ε, όπως φορά και την έρευνα για την πιθανή παρέμβαση στις εκλογές. Βεβαίω όλα αυτά δεν αφορούν άμεσα το θέμα μας, αλλά δείχνουν ότι υπάρχει ένα ανεπτυγμένο πλαίσιο ελέγχων. Τώρα για να επανέλθω στο πλαίσιο αυτό, η τελευταία εξέταση έδειξε ότι η ετήσια αυτή ε, εξέταση λειτουργία παίζει πλέον τον ρόλο της και γνωρίζουμε ε, το πώς πλέον λειτουργούν ή δεν λειτουργούν τα πράγματα στην πράξη και διαπιστώνουμε ότι σε κάποιες πτυχές απαιτείται περαιτέρω δουλειά για να υπάρξει αποτελεσματική προστασία. Άρα η έκθεση της Κομισιόν βλέπει ποια είναι τα περαιτέρω βήματα που πρέπει να γίνουν. Παραδείγματο χάρη το Συμβούλιο καταλήγει ότι ο τακτικό έλεγχο του Υπουργείου Εμπορίου πρέπει να εστιάσει περισσότερο σε ζητήματα που είναι σημαντικά, όπω η προστασία που ισχύει όταν διαβιβάζονται περαιτέρω τα δεδομένα αυτά που έχουν ληφθεί από την Ευρώπη επιπλέον. Ενώ η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου έχει εντείνει τι προσπαθίε της, θα πρέπει να μοιράζεται πληροφορίε. Ε, με την Κομισιόν για τις τρέχουσες έρευνες που κάνει και αυτό θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς συχνά εξετάζουμε παρόμοιες περιπτώσεις και πρακτικές. Για να καταλήξω λοιπόν, τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας ε, έχουμε δει σημαντική πρόοδο η εμπειρία μα με την καθημερινή λειτουργία του πλαισίου αυτού δείχνει επίση ε, τι περαιτέρω πτυχέ που μπορούν να βελτιωθούν και πρέπει να λάβουμε υπόψη πως ε, υπάρχουν υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του δικαστηρίου. Η άποψη τη ε, γενική Υγετρίας δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα. Θα πρέπει βεβαίω να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου για να δούμε τι ακριβώ αντίκτυπο θα έχει αυτή η υπόθεση σε διάφορα νομοθετήματα μεταξύ των οποίων και η ασπίδα αυτή προστασίας και βεβαίω ότι αποφασίσει το δικαστήριο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Να ευχαριστήσω λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας των Δεδομένων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σαφές ότι ο καθένας έχει τον ρόλο του και είναι διαφορετικός, οι απόψεις μας διαφέρουν. Ταυτόχρονα η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι μέσω της συνεργασίας έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε πραγματική πρόοδο προς όφελος των πολιτών στην εφαρμογή της ασπίδας αυτής αλλά και όσον αφορά το μοντέλο αυτό το οποίο αλλάζει στις ΕΠΑ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε κύριε Τσανκαρέλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και να ακούσουμε τώρα τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής για την προστασία των δεδομένων. Η κυρία Λίζα Μαρία Λάγκε, εκπρόσωπος ε, της αρχής της Γερμανικής για την προστασία δεδομένων και μετά τον κύριο Φρανσουά Πλερίνη από τη Γαλλική Σχετική Υπηρεσία. Έχετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί βουλευτές που μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το έργο μα για την ασπίδα προστασία τα τελευταία τρία χρόνια. Πρωτού περάσουμε στι λεπτομέρειε, να πω δύο λόγια για τη γενική αναθεώρηση και την εξέταση των, ε, της νομοθεσίας αυτής. Φέτος έχουμε από την Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία ε, και από την DPS ε, εκπροσώπους για να δείξουν τι γίνεται στην ασπίδα προστασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξετάζουμε από δύο διαφορετικές πλευρές την ασπίδα προστασίας. Κατά να έχει εφαρμοστεί το κείμενο όπως θα ε, πρέπει και εξετάζουμε και την, την ασπίδα προστασίας έχοντας υπόψη μας και όσα προβλέπει το GPDR και ο χάρτης των ελληνικών δικαιωμάτων καθώς και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που εκκρεμούν ακόμα. Θα κοιτάξουμε λοιπόν την ε, δομή της έκθεσης και θα σας δώσω μια παρουσίαση των βασικών εμβρημάτων από εμπορικής πλευράς και ο συνάδελφός μου μετά θα σας μιλήσει για την πρόσβαση των ε, δημοσίων αρχών σε ό,τι αφορά την ασπίδα προστασία. Από πλευρά εμπορική, η βασική ανησυχία είναι η έλλειψη βασική επισκόπηση και εφαρμογή. Κοίτατε τι σχετικέ δράσει, ε, κοιτάμε δράσει από το εμπορικά επιμελητήρια, από την ε, Ομοσπονδιακή το Υπουργείο Εμπορίου. Το Υπουργείο λοιπόν Εμπορίου έχει βελτιώσει την κατάσταση και τους ελέγχους ε, στα πλαίσια της, ε, του νόμου για τον ασφαλιλημένα. Επίσης, έχει αυξηθεί ε, ο, το ποσό των δημοτολεπτικών ελέγχων, των αυταπάγγελτων δημοτολεπτικών ελέγχων. Ωστόσο, επικεντρώνονται σε βασικά τυπικά στοιχεία κατά πόσον είναι πλήρε οι πολιτικέ, κατά πόσον υπάρχει σωστή διοργάνωση και κατά πόσον λειτουργούν οι σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα. Και το FGC λοιπόν έχει εστιαστεί πιο πολύ στις παραβιάσεις που αναφέρονται. Είναι πλέον στάνταρ διαδικασία να υπάρχει αναφορά στην Επιτροπή αυτή τέτοιων περιστατικών σε ό,τι αφορά εταιρείε οι οποίε έχουν παραβιάσει τι υπεσχέσει του σε ό,τι αφορά την ασπίδα προστασία. Ωστόσο, το FTC δεν μοιράστηκε μαζί μα τη στρατηγική υλοποίηση κατά τη διάρκεια τη αναθεώρησης. Επικεντρωνόμαστε και πάλι σε πιο τυπικά στοιχεία, κατά πόσο είναι έγκυρε, για παράδειγμα, διαδικασίες. Όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει ω τώρα δεν πηγαίνουν στην ουσία, δεν μπαίνουν στην ουσία. Αναλογικότητα, αναγκαιότητα των μέτρων. Δεν υπάρχουν λοιπόν ουσιαστικοί έλεγχοι για το τι συμβαίνει με τα δεδομένα τα οποία εμπίπτουν υπό την ασπίδα προστασίας. Δεν φαίνεται να υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες να οδηγούν σε τέτοιου ελέγχου και έτσι δεν ελέγχεται στην ουσία το όλο ζήτημα αυτό. Ένα τομέα ο οποίο επανειλημμένα επισημαίνεται είναι οι μεταφορέ. online. Είναι βασικό να υπάρχει προστασία των δεδομένων όπου και να μεταφέρονται τα δεδομένα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι η ασπίδα προστασίας και σε ό,τι αφορά τις ε, μεταφορές online υλοποιείται σωστά. Η ίδια η ασπίδα προστασίας, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά υπάρχει, είναι μηχανισμός αυτοπιστοποίησης, ε, σημαίνει ότι θα αποκαλύψουν, θα αποκαλύπτουν οι εταιρείε τι διατάξει του για των δεδομένων. Αυτό ακόμα δεν έχει συμβεί. Να δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, αξιότιμοι βουλευτέ. Θα σα αναφέρω τι γίνεται σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται στη ΣΥΠΑ υπό την ασπίδα προστασίας. Καταρχάς, το EDPB καλώς ορίζει τις σημαντικές βελτιώσεις που έγιναν από την τελευταία αναθεώρηση. Καταρχάς, ο διορισμός των τελευταίων ε, ε, μελών ε, του σχετικού σχετικής επιτροπής, μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά το σχέδιο εργασία και τον διορισμό του κυρίου Κιθ Κράκ, που είναι υφυπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ως μόνιμο διαμεσολαβητή από 18 Ιανουαρίου 2019. Ωστόσο, κάποια από τα βασικά σημεία που μας ανησυχούν και τα οποία υπήρχαν ήδη στις προηγούμενες εκθέσεις δεν έχουν ακόμα επιληθεί πλήρως. Σε ό,τι αφορά ανησυχίε για τέσσερα ζητήματα βασικά. Καταρχάς, τη διαδικασία συλλογή δεδομένων. Κατά δεύτερον, η επισκόπηση που υπάρχει στη διαδικασία αυτή. Κατά τρίτον, η ύπαρξη ε, σωστή ε, συλλογική ε, ε, συλλογικών εκδικάσεων και ο, ο μηχανισμός ε, προσφυγής. Αυτά τα τέσσερα θέματα λοιπόν θα κοιτάξουμε και τα σχετικά πορίσματα. Και μετά φυσικά θα είμαστε στην διάθεσή σας για ερωτήσεις. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα, συλλογή δεδομένων υπό διαφορετικά προγράμματα παρακολούθησης. Έχουμε διαφορετικά ζητήματα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και του τμήματος 702 και του 1203 ε, θεωρούμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη διαδικασία για να καθορίζεται κατά πόσον ένα άτομο ή κατά πόσον μια ομάδα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο παρακολούθησης και για καλύτερη παρακολούθηση των μεμονωμένων στόχων από ανεξάρτητες αρχές επειδή υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίε τις οποίες έχουμε τελικά πρόσβαση, δεν έχουμε δυνατότητα να αποκλείσουμε ότι υπάρχει μαζική και μη διακριτική πρόσβαση στο ό,τι αφορά το πλαίσιο του προγράμματος Upstream. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του 1203, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασία Δεδομένων θεωρούμε ότι ότι ενώ γίνονται τέτοιε μεταφορέ δεδομένων, οι διατάξεις του 1203 εμπίπτουν στο νομικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να αξιολογείται στα πλαίσια της ασπίδας προστασίας σε ό,τι αφορά τα στοιχεία τα οποία μας ε, προβλέπει η σχετική οδηγία DP-Date έχει πρέπει να σημαίνει ότι οι κανόνες αυτοί έχουν να κάνουν μόνο με την εκτελεστική οδηγία 1203 και όχι την 702 ε, του νόμου παρακολούθησης επικοινωνιών αλλοδαπών υπηρεσιών και πληροφοριών. Και η ομάδα παρακολούθησης εντόπισε δύο ζητήματα που μας ανησύχουν. Καταρχάς, το δεύτερο ε, τμήμα του 28 έχει να κάνει με την συλλογή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, Αυτές οι αναφορές που γίνονται στην υποσημείωση 5 έχουν να κάνουν και με έναν επιπλέον στόχο σε ό,τι αφορά τη συλλογή μυστικών ε, πληροφοριών για να είναι πιο εύκολη η στοχευμένη συλλογή δεδομένων. Από τις συζητήσεις με την εκπροσώπους του ΙΠΑ σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων, το Συμβούλιο για την ε, Προστασία των Δεδομένων κατανόησε ότι Πέρα από αυτά που προβλέπονται στα δεύτερη γενότητα, αν συλλέγονται τα δεδομένα αυτά, σκοπό έχουν να εντοπίσουν στοχευμένους ε, συγκεκριμένους στόχους. Αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει επιπλέον ε, προσπάθεια συλλογής δεδομένων και επειδή δεν μπορέσαμε να διευκρινίσουμε τι ακριβώς σημαίνει το προσωρινό αυτά, θα συνεχίσει η συλλογή δεδομένων έως ότου γίνει ταυτοποίηση του στόχου. Δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι παραβιάσεις της εγκληστικής οδηγίας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα δράση κατά ατόμων και κυρίω δεν μπορούν να σημαίνουν προσφυγή ότι θα καταγγελθούν τα άτομα αυτά στα δικαστηρία. Άλλο θέμα είναι το θέμα της επισκόπησης. Εντοπίζεται λοιπόν, διευκρινίζετε ότι υπάρχει σωστή δράση και ότι υπάρχουν ε, στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την ε, μυστικέ υπηρεσίε σε ό,τι αφορά τους ε, αξιωματούχους για, για θέματα ελευθερία και δυτική σφαίρα, την, Topic το Κογκρέσο και το Συντικό Δικαστήριο για την παρακολουθήση των επικοινωνιών. Αυτά έχουν να κάνουν με την έλλειψη πρόσβασης προϊόντων της διαδικασίας αυτής επιτήρησης. Επίσης, μία πιο λεπτομερής έκθεση για το πώς γίνονται εκατονεντές αυτές ε, οι διατάξεις στα προγράμματα ε, παρακολούθησης θα ήταν κάτι το ευπρόσδεκτο γιατί θα έδινε πιο πολλές πληροφορίες και θα διευκρίνιζαν όλες αυτές τις πτυχές και το ίδιο θα θέλαμε να γίνει και σε ό,τι το τμήμα 702 του ΦΙΖΑ, του νόμου ΦΙΖΑ για την παρακολουθήση επικοινωνιών αλλοδαπών υπηρεσιών και πληροφοριών. Και κάποιες ε, εκθέσεις οι οποίες δεν χορηγήθηκαν στην ομάδα για την ασπίδα προστασία, γιατί θεωρήθηκαν απόρριτε παρά το γεγονό ότι περιλαμβάνουν κρίσιμε πληροφορίε σε ό,τι αφορά τι ε, τρει εκθέσει του P-Club, οι οποίες ε, εκ των οποίων μία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Αυτές οι εκθέσεις λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντικές, γιατί η λειτουργία του νομοθετήματος αυτού δεν συζητήθηκε σε καμία περίπτωση στις προηγούμενες εκθέσεις. Και σε ό,τι αφορά τις γενικές ε, ανησυχίες για το θέμα αυτό, έχουμε να πούμε ότι η ομάδα παρακολούθησης ε, διατίθεται να εξετάσει υπέρτερο έγγραφα με φυσικά τη σχετική αν της επιτραπεί. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη συμφωνητή FTP. Και θεωρούμε ότι μια τέτοια πρόσβαση θα είχε αποτέλεσμα να έχουμε πιο σωστές ε, αξιολογήσεις. Το τρίτο θέμα. Το θέμα της... Μέτρων αποκατάστασης για ιδιωτών. Οι, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε προβλέπουν τέτοια μέτρα επανόρθωσης για τους ε, ε υπηκόους. Υπάρχει το σχετικό σχετική δράση για την αποκατάσταση και η ε, παρακολούθηση επικοινωνιών, το ΦΙΣΑ, παρακολούθηση επικοινωνιών αλλοδαπών υπηρεσιών πληροφοριών. Βέβαια, με βάση το φύσα ελάχιστε δυνατότητε δίνεται σε έναν υπηκό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να αμφισβητήσει την παρακολούθηση από διάφορε εταιρείε. Βέβαια, υπάρχει ε, το μόνιμο κριτήριο να ε, δοθούν αποδείξεις για το περιεχόμενο του κειμένου. Βέβαια, δεν είναι σίγουρο ότι πληρούνται δικονομικές ε, προϋποθέσεις από έναν ε, Ευρωπαίο υπήκο όταν υποβάλλει αγωγή με βάση το τμήμα νόμου 702 για την παρακολούθηση επικοινωνιών αλλοδαπών υπηρεσιών πληροφοριών. Το τέταρτο ζήτημα που θα ήθελα να σας αναφέρω αναφέρεται στο μηχανισμό του διαμεσολαβητή που θέλει να καλύψει κάποιες αβεβαιότητες για την πιθανότητα ε, ένας ε, Ευρωπαίος υπήκος να μπορεί να ε, γύρει αγωγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Βέβαια θα πρέπει να, γίνουν, να γίνει έλεγχος για ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσει. Τα δύο ζητήματα που αφορούν το ζήτημα αυτό είναι τα εξής. Ο μηχανισμός διαμεσολαβητή δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη. Το πρώτο αίτημα που υπευλήθη από Ευρωπαίο Υπήκο ήταν στα τέλη του 2018 και κρίθηκε μη παραδεκτή. Και ε, το δικό μας Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ε, θα αναθεωρήσει την, την όλη διαδικασία. Επίσης, εκφράζουμε την, ε, τις ανησυχίες μας για, τον, ε, για, την, για την ανεξαρτησία και το, τις αρμοδιότητες του διαμεσολαβητή, γιατί ο διαμεσολαβητής δεν έχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες και μπορούν ε, οι πληροφορίες να τροποποιηθούν από τους ε, επιθεωρητές ή τους βασικούς ανακριτές και ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί άμεσα να διορθώσει περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και ο διαμεσολαβητής ε, μπορεί να επισημάνει κάποιες παραβιάσεις του τμήματος 702 ή άλλης παραγράφου, αλλά δεν μπορεί να ε, εγείρει αγωγή ε, στο δικαστήριο, γιατί το δικαστήριο έχει διακριτική ευχαίρεια για το τι θα κάνει με τις πληροφορίες. Επίσης, ε, μπορεί να προταθεί δικαστική αναθεώρηση, και είναι δυνατόν να εγκριθούν κάποια μέτρα αποκατάστασης, εφόσον ο διαμεσολαβητής δεν δώσει απάντηση ή δώσει μη ικανοποιητική απάντηση προς τον ενάγοντα. Αυτά ως προς την τρίτη διαδικασία επανεξέτασης. Μάλιστα. Πριν ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να πω και εγώ λίγα λόγια και να επισημάνω ότι ο μηχανισμός αιτήσιας επανεξέτασης είναι πολύ χρήσιμος γιατί ε, μας κρατά συνέχεια σε εγρήγορση και μας για τους Αμερικανούς και δίνει κάποιες πιθανότητες ε, βελτίωσης. Ε, μάλιστα αποφασίσαμε να έχουμε πιο συχνές ε, συζητήσεις για κάποια κρεμή ζητήματα. Και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στα θέματα δεδομένων προσωπικού. Θα πρέπει και οι υπάλληλοι να έχουν την ίδια δυνατότητα πρόσβασης σε περίπτωση δεδομένων ανθρωπίνων πόρων. Μέχρι στιγμή πάντω ε, επαναλαμβάνω, το σε αιτήσει επανεξέταση απέδειξε ότι είναι πολύ χρήσιμο. Μάλιστα, ακούσαμε τους καλεσμένους μας και έχουμε χρόνο για συζήτηση. Θα πρότεινα λοιπόν οι συνάδελφοι θέλουν το λόγο να το δηλώσουν. Προηγούνται φυσικά οι συντονιστές. Εφόσον φυσικά ενδιαφέρονται να λάβουν το λόγο. Σίπελ, Ιντβελτ. Κυρία Σίπελ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους καλεσμένους για τις παρουσιάσεις τους. Και παρόλο που όλοι συμφωνούμε ότι έγιναν κάποιες βελτιώσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με τον ασφαλή λιμένα, ε, υπάρχουν κάποια ζητήματα που απορρέουν από τις τελευταίες, τις πιο πρόσφατες εκθέσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία ερώτηση για την εφαρμογή. Η έκθεση αναφέρει ε, μετά την ανάλυση δράσεων για τις 7 περιπτώσεις για την ασπίδα ιδιωτικότητας, ε, ε, επικρίνεται το περιορισμένο εύρος των πληροφοριών που σας έδωσαν. Τι γίνεται για να έχουμε πλήρη επισκόπηση της κατάστασης και την πιθανότητα υποβολής κυρώσεων και τι μπορούμε να κάνουμε για να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που δεν δίνουν οι Αμερικανοί. Σε ό,τι αφορά το μηχανισμό του διαμεσολαβητή, και το κατά πόσο είναι χρήσιμος ο μηχανισμός. Η έκθεση είναι σχετικά θετική για το διαμεσολαβήτη, αλλά ε, σε δύο περιπτώσεις ε, ο Γενικός Εισαγγελέας ε, έγειρε αμφιβολίες για την ομιμότητα αυτού του μηχανισμού διαμεσολάβησης, γιατί λέει ότι δεν δίνει, έχει ανεξαρτησίας ε, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα αμφισβήτησης τη αξιοπιστίας των δεδομένων ή της ε, καταγγελίας κάποιων παραβιάσεων ε, σε ό,τι αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες από τις υπηρεσίες πληροφοριών. Οπότε πώς συνδυάζονται όλα αυτά. Και η τελευταία ερώτηση αφορά τις εκκρεμωδικίες, ιδιαίτερα την περίπτωση SREMS 2. Από τη στιγμή που ε, εκδικάσεις αποφάσεις στο δικαστήριο, εκδικάσεις υποθέσεις στο δικαστήριο, ε, τι γίνεται με το διαμεσολαβητή. Ε, είπατε ότι είστε πολύ θετικοί για το μηχανισμό του διαμεσολαβητή, αλλά επειδή υπάρχει θέματα ε, ε μαζικής παρακολούθησης και το τρόπο που συγκεντρώνονται και δίνονται κάποια δεδομένα, θεωρείται ότι από τη στιγμή που υπάρχουν αμφιβολίες ε, από το δικαστήριο είναι όντως νόμιμη η ασπίδα ιδιωτικότητας, ε, μια και εσείς επιφυλαχθήκατε τις γνώμες σας να αναθεωρήσετε. Υπάρχουν ακόμη μαζικά δεδομένα. Οπότε υπάρχουν κάποιες ιδέες για να σταματήσει αυτή η μαζική συγκέντρωση δεδομένων. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Και αν όχι, υπάρχουν προτάσεις ή συμπληρωματική έλεγχη για να είμαστε σίγουροι ότι δεδομένα που δεν αφορούν συγκεκριμένη υπόθεση από τη στιγμή που θα μεταδοθούν τουλάχιστον θα διαγραφούν. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο για τις μελλοντικέ επανεξετάσεις αυτού του μέτρου. Ευχαριστώ. Μάλιστα, κυρία Ίντφελτ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας. Οι επανεξετάσεις αυτές είναι λίγο επαναληπτικές έως πολύ. Η Μπίρκετ Σίπελ ήταν ασυνήθιστα διπλωματική και επικής στα σχόλιά της. Διάβασα την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, άκουσα τις παρουσιάσεις σας, άκουσα και τον κύριο Τζανκαρέλη και διαρωτήθηκα. Για το ίδιο πρόγραμμα μιλάμε. Γιατί ανακεφαλαιώνοντας αυτά που είπατε εσείς και αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι η ασπίδα προστασίας ιδιωτικής σφαίρας είναι ανεπαρκής εγγύηση. Δεν εφαρμόζεται καλά, δεν ελέγχεται επαρκώς. Και ο κύριος Τζανκαρέλη είπε όλα είναι καλά. Αλληλούια. Χαιρόμαστε πολύ. Ε, από την ε, παρουσίαση του κυρίου Τζακαρέλη κρατήσαμε το χαρακτηρισμό επιτυχία, που σημαίνει ότι κατά τη γνώμη σας όλα βαίνουν καλώς με την ε, ασπίδα προστασίας. Και όταν λέω επαναληπτικές είναι οι συζητήσεις, γιατί το ίδιο είχαμε μια από τα ίδια και με το Safe Harbor. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ε, αποκρύψει, καταργήσει τις εκθέσεις ε, για το Safe Harbor γιατί το έκριναν πολύ αρνητικά και αποσιωπήθηκαν τελικά οι εκθέσεις. Να, αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν μας παίρνουν σοβαρά οι Ευρωπαίοι πολίτες γιατί εργαζόμαστε σκληρά, ε, νομοθετούμε, εργάζεται σκληρά ο κ. Τζανκαρέλη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και μετά τα καταπατούμε όλα μετά από ένα αίτημα των ε, Ηνωμένων Πολιτειών και μετά ε, τους θερμοπαρακαλούμε ε, μήπως θα μπορούσαν, μήπως είχα την καλοσύνη να εφαρμόσουν έστω και λίγα από αυτά που συμφωνήσαμε. Είναι ε, ανεπαρκείς οι αρμοδιότητες και εξουσίες του διαμεσολαβητή λόγω της επέμβασης του Τραμπ. Μα είμαστε σοβαροί. Πώς θα το παρουσιάσουμε αυτό και θα το εξηγήσουμε στους ε, ψηφοφόρους μας. Δεν θα έχουμε τα, το τη δυνατότητα. Είναι ε, σαν φιλοσικής αυτή η ασπίδα ασφαλεία. Καλύτερα έτσι να ονομάσουμε. Φιλοσικής για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας. Και με προβληματίζει και ο τρόπος που το χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, γιατί φαίνεται ότι διαπραγματεύεστε μία συμφωνία με τους Αμερικανούς για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Οπότε και εκεί με τα φίδια. Γιατί Μπορεί να κάνουμε συμφωνίες, αλλά εφαρμόζονται. Μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα εξασφαλίσει εφαρμογή τους, γιατί θα έρθει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μας ζητήσει τη συνένεσή μας για τις, για τις συμφωνίες αυτές. Και αν κρίνω την αξιοπιστία της ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον τρόπο που χειρίζεται το Safe Harbor και την ασπίδα προστασία ιδιωτικότητα, εγώ δεν βρίσκω κανένα λόγο να δώσουμε τη συγκατάθεσή μα για οποιαδήποτε άλλη παρόμοια συμφωνία. Πραγματικά έχω α, κουραστεί, γιατί κάθε χρόνο μία από τα ίδια α, ακούμε. Δεν λειτουργεί η συμφωνία, ανεπαρκής, δεν εφαρμόζεται σωστά ή εφαρμόζεται πλημελώς. Ε, μην μας κουράζετε κάθε χρόνο με τα ίδια και τα ίδια κάνετε κάτι διαφορετικό. Θα έλεγα να ολοκληρώσουμε το γύρο των αγορητών και μετά να δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας για να απαντήσουν στις απορίες των Ευρωβουλευτών. Και πριν να ολοκληρώσουμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Φως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τα μέλη του πάνελ. Να άκουσα και τους τρεις και νομίζω έτσι πως η έκθεση έχει μια αρκετά καλή βάση αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Και εδώ έχω πάντα την αίσθηση πως είμαστε σε καλό δρόμο. Ο κ. Σικαρέλη μας είπε «Ε, διαβίβαση δεδομένων, καλύτερη ανταλλαγή, εφαρμογή του δικαίου. Το ερώτημά μου είναι υπάρχουν κάποιες άλλες ιδέες ή κάποια άλλη προσέγγιση που διαπραγματεύεστε με την Αμερικανική πλευρά για την βελτίωση με τα κυρία Λάγκε μια ερώτηση για εσάς ε, αν κατάλαβα καλά στην εφαρμογή της ασπίδας αυτής από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου δεν εξετάζεται το τι γίνονται τα δεδομένα. Έτσι κατάλαβα εγώ τουλάχιστον. Θα ήθελα να γνωρίζω τι κάνετε λοιπόν εσείς εδώ που δεν κάνουν εκεί. Για να έχουμε έτσι μια ιδέα του τι γίνεται, τι λείπει και τι επιπτώσεις έχει αυτό. Και κύριε Πελεγκρίνη, εσείς περιοριστήκατε στις εξελίξεις γύρω από το θέμα της Φάιζα ε, στα τρία από τα τέσσερα κεφάλαια στα οποία αναφερθήκατε δηλαδή και σε σχέση με τον ε, επόπτη είπατε ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται ακόμα γιατί κανείς ακόμα δεν έχει υποβάλει κάποια καταγγελία. Αν λοιπόν υπήρχε μια τέτοια καταγγελία θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, θα είχατε κάνει κάτι. Σας ευχαριστώ κύριε Κόρνερ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτά τα οποία είπατε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του Facebook. Εδώ πέρα αναφέρεται ότι υπάρχει ξεκάθαρη ευθύνη και πρέπει να σταματήσει η μεταφορά των δεδομένων. Μετά ε, ειδικά αν δεν έχουν τηρηθεί τα όσα ορίζει η νομοθεσία σε σχέση με τη μεταφορά δεδομένων το, στη ΣΥΠΑ. Αυτή είναι η άποψη του Γενικού Εισαγγελέα. Και μετά, από τη σελίδα 55 ως 59, ο Γενικός Εισαγγελέας αναλύει το γιατί η ασπίδα ιδιωτικότητας είναι μόνο στα χαρτιά και δεν εγγυάται πλήρως στην ιδιωτική σφαίρα. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής πρέπει στο μέλλον, εάν αποφασίσει το δικαστήριο σχετικά, να υπάρξει απαγόρευση της μεταφοράς δεδομένων σε τρίτες χώρες όπου υπάρχει μαζική παρακολούθηση όπως ε, από ό,τι φαίνεται γίνεται από όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις των ΗΠΑ και δεύτερον είναι σαφές τώρα το ότι η ασπίδα αυτή παραπέει ε, δεν νομίζω να υπάρξει κάποια επανεξέταση αν δούμε την υπόθεση ΣΡΕΜΣ όπου ο Γενικός λέει εντάξει είμαι κατά αλλά να το δούμε αν δεν γίνει τώρα θα γίνει στην επόμενη υπόθεση τι κάνει η Κομισιόν, τι θα κάνετε στο μέλλον γι' αυτό και τελευταία ερώτηση επικεντρωνόμαστε στις ΙΠΑ αλλά αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι οι εξελίξεις στην Κίνα Έχουμε όλο και περισσότερες ε, ε, επιχειρήσεις. Θα αναφέρω μόνο το TikTok, που εκατομμύρια έφηβοι ανεβάζουν τα δεδομένα τους ε, και τα βλέπουν οι κινέζικες αρχές ασφαλείας. Τι κάνει εκεί πέρα η Κομισιόν συγκεκριμένα για την προστασία των δεδομένων των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ κύριε Μπράιρ, έχετε τον λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων για την δουλειά που κάνετε στο ζήτημα αυτό. Εγώ πάντα έλεγα ότι ε, πρόκειται για μια φάρσα και δεν αξίζει το όνομα ασπίδα προστασίας δεδομένων γιατί δεν αντιμετωπίζει τις ελλείψεις και του προηγούμενου καθεστώτος, δηλαδή δεν μας προστατεύει από την μαζική παρακολούθηση την οποία αποκάλυψε ο Έντουαρτ Σνόντεν. Και η άποψη του Γενικού Εισαγγελέα έχει έκθεσή τις διάφορες ελλείψεις ε, της απόφασης αυτής, αλλά θα ήθελα να τονίσω το ότι τα κράτη-μέλη ε, είναι υπεύθυνα για την εθνική ασφάλεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα όσα κάνουν οι ΙΠΑ ε, υπό το πρίσμα αυτό δεν μπορούν να εξεταστούν. στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και δεν μπορούν να εξεταστούν όταν αποφασίζουμε για την επάρκεια άλλων κρατών και κυβερνήσεων. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, αλλά και το θέμα της παραβίασης ανθρωπινών δικαιωμάτων στη χρήση των δεδομένων αυτών στον πόλεμο κατά της δημοκρατίας που οδήγησε σε κρατήσεις, ε, λίστες απαγόρευσης πτήσεων, ε, απαγωγές κτλ. Και ήδη αναφερθήκατε στο θέμα της προσφυγής στα δικαστήρια, αλλά ακόμα και οι λίγε προστασίε που υπάρχουν δεν μπορούν να επιβληθούν σε ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι και θέμα του ότι η Αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να επικαλεστεί το ότι κάποια δεδομένα είναι απόρριτα και δεν μπορούν να ακουστούν σε δικαστήριο γιατί κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια. Κάτι το οποίο έχει γίνει επανειλημμένως. Τώρα, η προτινόμενη λύση δηλαδή ότι θα πρέπει οι αρχές προστασίας δεδομένων να σταματήσουν ατομικά την ροή δεδομένων που επηρεάζονται από αυτές τις ελλείψεις είναι μη ρεαλιστική γιατί όλες οι ροές δεδομένων επηρεάζονται από αυτές τις ελλείψεις και άρα ελπίζω το δικαστήριο να ακυρώσει αυτό το καθώς. Έχω μία ερώτηση προς την Κομισιόν. Εάν το δικαστήριο ακυρώσει την ασπίδα αυτή, έχουν υπάρξει απόπειρες ε, στη ΣΥΠΑ να υπάρξει κάποια προσφυγή στα δικαστήρια γι' αυτό το ζήτημα, ειδικά στην ε, Καλιφόρνια, όπου βασίζονται πολλές από αυτές τις εταιρείες. Εάν κάποιο, κάποια Αμερικανική πολιτεία, όπως η Καλιφόρνια, ε, αποφασίσει να ζητήσει μία απόφαση επάρκειας, θα το εξετάσει η Κομισιόν, μπορεί μία μεμονωμένη πολιτεία να κάνει μία τέτοια αίτηση. Να σα υπενθυμίσω, Λίγο ο ότι το επόμενο θέμα, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διατάξη έχει μείνει αναβληθεί, αλλά μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τι 12 είχαμε χρόνο για το θέμα αυτό. Προφανώ θα ξεπεράσουμε το χρόνο που έχει προβλεφθεί, αλλά να το έχετε παρακαλώ υπόψη σας όταν κάνετε ερωτήσεις. Για να έχουν χρόνο να απαντήσουν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω και τους ομιλητές που ήρθαν εδώ. Προσπαθώ να καταλάβω το σενάριο αυτό. Από τη μία έχουμε ε, επανειλημμένα θέματα που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άρα έχουμε θέματα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασία Δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασία Δεδομένων. Όλοι θέτουν σημαντικά ζητήματα σε ό,τι αφορά την ασπίδα προστασία και μετά έχουμε και την άλλη πλευρά που λέει άλλα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι γίνεται και πώς μπορείτε να λέτε ότι όλα πάνε καλά, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις μεν. Είναι λες και βάφουμε έναν εξωτερικό τοίχο ενός σπιτιού και ξέρουμε ότι μέσα τα θεμέλια είναι σαθρά. Αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι οι δικλείδες ασφαλείας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του νόμου και θέματα εθνικής ασφάλειας. Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσον έχει σταματήσει η Αμερική να κάνει τέτοια μαζική συλλογή δεδομένων. Αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι μάλλον έχει σταματήσει βάσει αυτά που λένε οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ που ενδεχομένω να ψεύδονται για οικονομικά τέτοια συμφέροντα και να κρύβουν αυτά που συμβαίνουν. Και η έκθεση σας αναφέρει και λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν επιλογής αυτό λέει η έκθεση. Και να πιστεύουμε ότι πλέον ε, τα δεδομένα αυτά είναι στοχευμένα, δεν ε, ε, συλλέγονται μαζικά. Δεν λέτε όμως ότι μας έχουν πει κάτι τέτοιο. Υπάρχει η ευρεία αυτή η πρόσβαση την οποία την παρακολουθούν κάποιοι αναλυτέ, αλλά δεν υπάρχει οποιαδήποτε δίκλυδα ασφαλεία ότι οι μέθοδοι για την πρόσβαση στα δεδομένα έχουν επιλεχθεί. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το πώ αποθηκεύονται, πώ συλλέγονται τα στοιχεία αυτά και το καθεξής. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η κατάσταση η οποία αντιμετωπίζεται. Είναι η εξή. Έχουμε οργανώσει που έχουν αποδεχτεί ότι λένε ψέματα και η νομοθεσία έχει αποδεχτεί ανεπαρκής. Πώς την εμπιστευόμαστε λοιπόν. Ανησυχώ λοιπόν και θα συμφωνήσω με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι για το μηχανισμό εποπτείας. Μιλάμε για έναν εξάρτητο διαμεσολαβητή, αλλά μιλάμε και για μέλος ε, του, Υπουργείου, του Αμερικανικού Υπουργείου. Ένα δικαστήριο εποπτείας ε, που εφαρμόζει ένα νόμο ο οποίος προβλέπει το απόρριτο. Άρα ο μηχανισμός αυτός εποπτείας βασίζεται σε μη διαφανείς ε, πληροφορίες οι οποίες είναι εντελώς ανεπαρκείς. Δεν ε, καταλαβαίνω τι γίνεται και να πω και το κάτι άλλο. Αν ε, τεθεί εκτός λειτουργίας η προστασία, τι θα γίνει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Να δώσουμε το λόγο λοιπόν στους προσκεκλημένους μας για να απαντήσουν. Από ό,τι βλέπετε υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε ό,τι αφορά τις εξέλιξεις για την ασπίδα προστασίας. Ο κ. Τζανκαρέλη έχει πάλι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις. Να ξεκινήσουμε μια περιπλοκή ερώτηση. Με ένα ναι σε ό,τι αφορά το θέμα της Καλιφόρνιας η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, ο κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, προβλέπει την δυνατότητα να υπάρχει σωστή αναγνώριση. Ότι αφορά την Αμερική επάρκεια και αυτό γίνεται σε επίπεδο των πολιτιών γιατί στον GDPR είχαμε προβλέψει το γεγονός ότι κάποια ομοσπονδιακά ε, συστήματα, κάποιες πολιτείες ενδεχομένως για κάποιους λόγους να αποφάσιζαν να εφαρμόσουν ε, ε, νομοθεσία για την ιδιωτική ζωή. Η διαδικασία λοιπόν συνεχίζεται σε ό,τι αφορά την Καλιφόρνια. Είναι ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε, να δούμε τι νέε ιδέε κατατίθενται. Η απάντηση λοιπόν είναι ναι, ε, φυσικά βέβαια εξαρτάται και το, από το τι θα αποφασιστεί στην Καλιφόρνια, ποια θα είναι η νομοθεσία και κατά πόσο θα πληρεί τις προδιαγραφές. Αυτό με οδηγεί και σε ένα άλλο θέμα. Αυτή είναι η λύση στη τελική ανάλυση. Αν θέλουμε να υπάρχουν μακροπρόθεσμα κάποια σωστή λύση, θα πρέπει να βασίζεται σε συντάγματα, σε νομοθεσία, η οποία θα πρέπει να είναι όσο πιο ευρεία γίνεται. Ακούσαμε να υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ σας, αλλά για ένα πράγμα συμφωνούμε. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε προς τους Αμερικανούς ομολόγους με τα μέλη του Κογκρέσου. Και γι' αυτό είναι και τόσο σημαντική η δουλειά που γίνεται για ένα νόμο σε ομοσπονδιακό επίπεδο στην Αμερική. Να δω τις άλλες ερωτήσεις, καταρχάς από την κυρία Σίπελ για το τι εννοούμε σε ό,τι αφορά το σκέλος της ε, ε, υλοποίησης της εφαρμογής. Έχουμε πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις δράσεις, τις μελέτες, τις έρευνες που γίνονται και που έχουν ολοκληρωθεί μάλιστα. Υπήρξαν κυρώσεις ε, και είδαμε εταιρείε οι οποίες ψευδώς ισχυρίστηκαν ότι συμμορφώνονταν με την ασπίτα προστασίας. Αυτό που τονίζουμε στην έκθεση είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις ε, δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για έρευνες εν εξελίξη. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πιο γρήγορες έρευνες είναι οι πιο κλασικές, αν θέλετε, έρευνες, ή τα πιο κλασικά ζητήματα, όπως είπαν και οι συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, είναι οι πιο εύκολες αυτές οι ε, υποθέσεις. όπου γίνεται γρήγορα, γρήγορα μία τέτοια έρευνα η οποία κλείνει και γρήγορα. Οι πιο περίπλοκες ε, έρευνες και αυτές που αγγίζουν θέματα ουσίας είναι αυτές που έχουν την πιο μεγάλη σημασία. Και εδώ έχουμε δει πιο πολύ εξέλιξη από πλευρά των ΙΠΑ. Και περιμένουμε λοιπόν μεγάλες αποφάσεις σε ό,τι αφορά τη Facebook και άλλες τέτοιε μεγάλες υποθέσεις. Και πολύ απλά θεωρούμε ότι μιας και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού η δυνάμεις, η τα, τα Συμβούλια Προστασίας Δεδομένων και η Επιτροπή Εμπορίου και άλλες αρχές, αλλά εν πάση περιπτώσει, ερευνούν τις ίδιες πρακτικές εκ παραλλήλου, θα υπήρχε μεγάλο όφελος για την ανταλλαγή, από την ανταλλαγή ε, πληροφοριών κατά τη διάρκεια των ερευνών θα διευκόλυνε τα πράγματα και από τις δύο πλευρές. Αυτό προσπαθούμε λοιπόν να λέμε ότι Καλό είναι να είμαστε ενημερωμένοι εκ των υστέρων, αλλά η ασπίδα προστασία προβλέπει και μια διαρκή ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσει, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μιας αποτελεσματική συνεργασία και των δύο πλευρών. Ελπίζω έτσι να διευκρινίζω λοιπόν το τι εννοούσα και ζητώ συγγνώμη αν δεν ήταν σαφέ εξ αρχής. Μου λέτε στη συνέχεια ότι άλλα λέτε και άλλα συμβαίνουν. Δεν λέω αλληλούια, αλλά πραγματικά κάποια πράγματα λειτουργούν. Λειτουργούν καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Και χαίρομαι που μα λέει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασία Δεδομένων ότι θεωρούν ότι αυτή η άσκηση δεν είναι μονοτυπική, έχει και ουσιαστικό όφελο. Εκ παραλλήλου, διαπιστώνουμε ότι ενδεχομένω να χρειαστεί να εργαστούμε περαιτέρω σε όλα αυτά μετά και από τι δικαστικέ αποφάσει. Επαναλαμβάνω, αυτό θα έλεγα και για οποιαδήποτε δικαστική εκδίκαση. Όσο περιμένουμε απόφαση δικαστηρίου, δεν μπορούμε να εικάζουμε το τι θα συμβεί. και κατά πόσον η δικαστική απόφαση θα σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Αν αυτή είναι η εντολή μας θα το κάνουμε. Αλλά αυτό ισχύει για όλες τις δικαστικές υποθέσεις και σημειώνω ότι ότι η γνωμοδότηση, η έκθεση περιλαμβάνει και κάποιες ε, σημαντικές εξέλιξεις για την ασπίδα, αλλά η γνωμοδότηση περιλαμβάνει επίσης ότι κατά τη γνώμη του εισαγγελέα η ασπίδα προστασίας δεν ε, σχετίζεται, δεν έχει σημασία για την προκειμένη υπόθεση που έχει να κάνει ε, πιο πολύ με βασικές διατάξεις και τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Αυτό λοιπόν. Και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι συμμετέχει στην προκειμένη περίπτωση. Για την Επιτροπή, συγγνώμη. Και αυτό με οδηγεί σε ένα άλλο θέμα, σε ό,τι αφορά την Κίνα, σε ό,τι αφορά τις μεταφορές οι μεταφορές αυτές προς την, από την Κίνα δεν βασίζονται σε οποιαδήποτε τέτοια απόφαση. Γιατί προφανώς η χώρα αυτή δεν θα πληρούσε τους σχετικούς όρους. Άρα υπάρχει το θέμα της παραβίασης των υποποιημένων συμβατικών ρήτρων. Και αυτό τονίζεται στην ομοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα. Επίσης, ετέθησαν ε, ερωτήματα για τον ε, διαμεσολαβητή και για την μαζική συλλογή δεδομένων. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τον διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής. Εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Δεν είναι σε καμία περίπτωση η μοναδική πηγή και η μοναδική λύση για προσφυγή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση του κοινού για θέματα εθνικής ασφάλειας. Υπάρχουν κι άλλα, κι άλλοι οδοί, οι δικαστικές οδοί, όπως και το δικό μας εσωτερικό σύστημα, διοικητικές διαδικασίε και του καθεξής. Έχουμε διαπιστώσει ότι όντως ο πύχης είναι αρκετά υψηλός, όπως και στο δικό μας το σύστημα. Και άρα, για να διευκολυνθεί η δυνατότητα που έχουν οι πολίτες να προσφεύγουν, έχουμε προσθέσει επιπροσθέτως το μηχανισμό του διαμεσολαβητή για να υπάρχει άλλη μια δυνατότητα προσφυγής πέρα από τις ε, εφιστάμενες. Και αυτό που προσπάθησα σήμερα να εξηγήσω είναι το εξή. Ο διαμεσολαβητής δεν είναι μόνος του, δεν εργάζεται μόνος του. Όταν κάνει μια έρευνα ο διαμεσολαβητής όταν λαμβάνει μια απόφαση. Και αν του ζητηθεί να προβεί σε διορθωτικά μέτρα, συνεργάζεται με απόλυτα ανεξάρτητες αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών αρχών. Δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι ο Γενικός επιθερητής των Μυστικών Πληροφοριών, ο οποίος ε, ήταν και αυτός που ξεκίνησε την παραπομπή του Προέδρου των ΗΠΑ, δεν είναι ανεξάρτητη μορφή που έχει και σημαντική εξουσία. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν στοιχείο το οποίο έχει να κάνει με την μηχανισμό α, του Μεσολαβητή και σε ό,τι αφορά την ομάδα του ΦΑΙΖΑ, του νόμου παρακολούθησης επικοινωνιών αλλά υπηρεσιών πληροφοριών. Επίσης και ο επικεφαλής μπορεί να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις και να ζητήσει διόρθωση τέτοιων παραβιάσεων, να διαγραφούν δηλαδή τα δεδομένα τα οποία ε, συλλέχθησαν παράνομα. Υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι δυνατότητες. Ξέρω ότι έχετε διαφορετικές απόψεις για τον διαμεσολαβητή, αλλά να το λάβετε και αυτό υπόψη σε κάθε περίπτωση. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία τώρα του διαμεσολαβητή, και με τα άλλα αυτά σώματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του μηχανισμού των είπα. Και αυτό το επιβεβαιώνει η αιτήσια επανεξετάση. Και για το θέμα της μαζικής παρακολούθησης, ε, συγκέντρωσης μάλλον δεδομένων, θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο και να σας τα εξηγήσει πιο διεξοδικά. Ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε για την οργάνωση αυτής της συζήτησης. Σε ό,τι αφορά τη μαζική συγκέντρωση δεδομένων, το σημείο αφετηρίας είναι ότι στις Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχει ε, ένας ε, νόμος του, της που λέει ε, πώς θα συγκεντρώνονται τέτοια στοιχεία. Πρόκειται για το νόμο ΦΙΣΑ που αποκλεί τέτοια συγκέντρωση, μαζική συγκέντρωση δεδομένων. Και αυτό το έχουμε αναφέρει και σε εκθέσεις μας, αλλά καλό είναι να το έχουμε υπόψη. Ο νόμος ΦΙΣΑ αποκλείει τη μαζική συγκέντρωση δεδομένων για την παρακολούθηση ε, αλλοδαπών υπηρεσιών πληροφοριών εντός των ΗΠΑ. Σε ό,τι αφορά την ανεπάρκεια, όταν έχουν σταλεί δεδομένα στις ΗΠΑ και τα κρατά ένα πάροχο υπηρεσιών, αποκλείεται δια νόμου ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες η μαζική συγκέντρωση δεδομένων. Και ο νόμος ΦΙΣΑ και το τμήμα 702 του νόμου ΦΙΣΑ, που συνήθως είναι το τμήμα που εγείρει τις περισσότερες ανησυχίες και είναι και η βάση για, τον, για το πρόγραμμα Upstream και το πρίσμα, απαιτεί στοχευμένη συγκέντρωση δεδομένων αυτό το τμήμα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει συγκέντρωση μόνο βάσει των επιλογέων. Και ο επιλογέας είναι μια δυνατότητα επικοινωνία, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και δεν είναι γενική όρη επιλογής βόμβα, τρόμος κτλ. Πρόκειται για μια διευκόλυνση επικοινωνία, όπως μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακόμη και με το τμήμα 702, δεν προβλέπεται εξατομικευμένος έλεγχος του δικαστηρίου για την επιλογή των επιλογέων. Παρ' αυτά, το δικαστήριο εκ των προτέρων ε, εγκρίνει τις διαδικασίες ε, στόχευσης και αυτές οι διαδικασίες στόχευσης λαμβάνουν υπόψη διάφορα στοιχεία για το πώς οι μυστικές υπηρεσίες όπως η NSA, η ESA, το FBI, CIA, η FBI μπορούν να επιλέξουν τον επιλογέα. Και με ποιες ενδείξεις ε, θα πρέπει μια τέτοια μυστική υπηρεσία να επιλέγει τον επιλογέα. Δεν είναι θέματα δηλαδή διακριτικής ε, είναι θέμα διακριτικής ευχαίρειας των μυστικών υπηρεσιών, αλλά το δικαστήριο εκ των προτέρων ε, εγκρίνει αυτές τις διαδικασίες στόχευσης. Και αυτό φαίνεται και στην έκθεση του P-Club, που είναι η αποπτικός φορέας για τις πολιτικές ελευθερίες. Και η έκθεση αυτού του P-Club είναι σημαντικό στοιχείο της ανεξάρτητης δομής εποπτείας των Πολιτειών και ε, έχει ε, ελεγχθεί το τμήμα 702 του νόμου ΦΙΣΑ. Και μάλιστα η έκθεση αυτή είναι 700 σελίδων και έχει στηριχθεί σε εμπιστευτικές πληροφορίες, σε απόρριτες πληροφορίες, οποίες εμείς δεν έχουμε πρόσβαση καμία και ευλόγος. Αλλά το P-Club έχει λάβει όλες αυτές τις απόρριτες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ και έχει συντάξει μια έκθεση στην οποία αποφαίνεται το τμήμα 702 αφορά στοχευμένη συγκέντρωση πληροφοριών και όχι μαζική και είναι αναλογική εφαρμογή του. Και με εκπλήσει που οι συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητούν ζητά νέα έκθεση γιατί θεωρεί ότι έχουν γίνει σημαντικές τροπολογίες στο ΦΙΣΑ. Όντως έχει εγκριθεί το ΦΙΣΑ, αλλά όλες οι τροπολογίες βελτιώνουν την προστασία της ιδιωτικότητας σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο του ΦΙΣΑ. Και για το τμήμα 702 δεν έχει γίνει καμία αλλαγή. Και πριν από δύο χρόνια το P-Club ε, μια έκθεση που εξακολουθεί να είναι έγκυρη και ενισχύει μια και δεν ε, έχει επηρεαστεί το πόρισμα της από τις αλλαγές που έχουν γίνει σχετική νομοθεσία. Πάντως και οι δικές μας χώρες μέλη κάνουν διάκριση μεταξύ της συγκέντρωσης δεδομένων εντός και εκτός επικράτειάς μας. Και ο νόμος ΦΙΣΑ, περί παρακολούθηση επικοινωνιών αλλοδαπών ε, μυστικών υπηρεσιών, ακόμη και εκεί και πέραν του τι σημαίνει ε, πόρισμα επάρκειας, λαμβάνεται υπόψη το πεδίο εφαρμογή. Πάντως αναλύσαμε την εκτελεστική εντολή και ακόμη και εκεί δεν έχουμε μαζική παρακολούθηση. Μπορούμε να έχουμε κατεξαίρεση μαζική συλλογή δεδομένων, αλλά με βάση την οδηγία 28, την προεδρική οδηγία πολιτικής 28, έχουμε λάβει διασφαλίσεις και διαβεβαιώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Διευθυντή ε, ε, Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που εποπτεύει τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ έχουμε λάβει τις διαβεβαιώσεις ότι γίνεται κατά ε, μαζική συγκέντρωση πληροφοριών και λαμβάνεται υπόψη η ασπίδα προστασίας στην έκτακτη αυτή συγκέντρωση, μαζική συγκέντρωση πληροφοριών. Κάποιος ευρωβουλευτής είπε ότι η μαζική συγκέντρωση δεδομένων απαγορεύεται ολοσχερώς από το ενωσιακό δίκαιο. Δεν ισχύει αυτό όμως. Αν δείτε την ομολογία του ΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ομολογία προβλέπει ότι η μαζική συγκέντρωση δεδομένων δεν απαγορεύεται ε, επιτρέπεται υπό όρους και με ασφαλιστικές δικλίδες. Το δικαστήριο έχει πει ότι γενικευμένη πρόσβαση σε περιεχόμενο απαγορεύεται. Αλλά αυτό α, μαζική παρακολούθηση και όχι μαζική συγκέντρωση δεδομένων. Και η γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα επιβεβαιώνει ότι η μαζική συγκέντρωση δεδομένων μπορεί να επιτρέπεται εφόσον χρησιμοποιείται για τη φιλτράρισμα στοχευμένων πληροφοριών. Και αυτό είναι μαζική παρακολούθηση. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη ότι και τα κράτη-μέλη επιτρέπουν μερικές φορές μαζική συγκέντρωση δεδομένων. Και έχει φανεί και σε μία μελέτη. Στο, το γερμανικό δίκαιο επιτρέπει ε, συλλογή μέχρι 30% των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οπότε υπάρχει αυτή η μαζική ε, συγκέντρωση δεδομένων και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν απαγορεύεται λοιπόν και δεν μπορούμε να πούμε ότι απαγορεύεται για μια ξένη χώρα. Και εφαρμόζεται αυτή η μαζική συγκέντρωση και από τα κρατη γιατί μερικέ φορέ χρειάζεται. Δεν λέω ότι θα πρέπει να είναι ο κανόνα. Εξαίρεση θα πρέπει να είναι και θα πρέπει να συνοδεύεται από ασφαλιστικέ δικλείδε και από εχέγγυα. Αυτό λέει και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Επίση και το Δικαστήριο του Στρασβούργου δίνει κάποια διακριτική ευχαίρεια στα κρατη για να χειρίσουν το ζήτημα αυτό τη μαζική συγκέντρωση δεδομένων. Οπότε θεωρούμε ότι κάτι αντίστοιχο πρέπει να ισχύει και για τρίτη χώρα όταν αξιολογούμε την επάρκειά της. Πάντως στις Ηνωμένε Πολιτείε δια νόμου απαγορεύεται η μαζική συγκέντρωση δεδομένων και μόνο εκτάκτως λαμβάνει η χώρα εκτός των Ηνωμένων Πολιτείων σε περίπτωση που τα δεδομένα μεταφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Μα έχετε μιλήσει για ένα 20 λεπτό και παραπάνω. Ξέρω ότι είναι περίμαχα αυτά τα θέματα και πολλές ερωτήσεις ε, στράφηκαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έχουμε και άλλου δύο καλεσμένους, δεν μπορείτε να μονοπολείτε την απάντηση. Και παρακαλώ δείξτε μία αυτοσυγκράτηση στην ε, ομιλία σας, στην ε, χρήση του, όρου, του χρόνου Ομιλία. Παρακαλώ. Περισσότερε ερωτήσει βέβαια αποτάθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ίσω και εσεί θέλετε το λόγο για κάποια σχόλια. Προσπαθήστε όμως να είστε πιο συνοπτικός, πιο λακωνικός από τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντιλαμβάνομαι βέβαια, αντιλαμβάνομαι και εκτιμώ ε, ιδιαίτερος την κατανόηση που θα δείξετε στη διαχείριση του χρόνου ομιλίας γιατί έχουμε μία μερή σε διάταξη και συνηθίζουμε να υπερβαίνουμε το ωράριό μας, αλλά να μην το παρακάνουμε κιόλα. Ask in German, I would like to answer in German. Μια που με ρωτήσατε στα γερμανικά, θα ήθελα να απαντήσω στα γερμανικά, κύριε Φως. Με ρωτήσατε πώς ερευνούμε το τι συμβαίνει με τα δεδομένα στην Ευρώπη όταν ασκούμε κριτική στη ΣΥΠΑ. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα κουλτούρας και πολύ διαφορετικό. Στην Ευρώπη έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες, οπότε οι εταιρείε υπολογίζουν ότι θα έχουν μια εταιρεία, μια αρχή η οποία θα υποπτεύει αυτά τα ζητήματα, οπότε υπάρχει ήδη αυτή η κουλτούρα, αλλά όσον αφορά τις ε, διεθνείς μεταφορές δεδομένων, ε, κατ' ουσίαν δεν υπάρχουν σχεδόν ποτέ ε, καταγγελίες γιατί πρώτα απ' όλα πώς το διαπιστώνει κανείς ότι έχουν μεταφερθεί διεθνώς τα δεδομένα του οπότε υπάρχει ανάγκη να γνωρίζουμε πρώτα απ' όλα ότι έχει υπάρξει μια τέτοια μεταφορά επιπλέον ε, αυτό είναι μια είναι το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων όπου έπρεπε να συμβιβαστούν η ευρωπαϊκή και η αμερικανική αντίληψη Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να φροντίσουμε ε, πρώτα απ' όλα να εννοούμε το ίδιο πράγμα όταν λέμε κάτι και με κάποιον τρόπο πρέπει να γίνει αυτό. Και βεβαίως ε, όταν μιλάμε για ένα μηχανισμό αυτοπιστοποίησης ε, αυτό δεν λαμβάνει χώρα αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο για να διασφαλίσουμε ότι όταν έχουμε το ίδιο κείμενο μπροστά μας εννοούμε τα ίδια πράγματα. Κύριε Πελεγρίνη, και παρακαλώ να είστε σύντομος. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Βοσ. Δεν μιλήσαμε μόνο για την ε, Φάιζα, γιατί η Φάιζα αφορά την στοχευμένη συλλογή σε αμερικανικό έδαφος ενώ εμείς λέμε ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες εκτός αμερικανικής επικράτειας, ειδικά η κυκλοφορία δεδομένων προς τις ΗΠΑ, θα πρέπει επίσης να καλύπτεται, να καλύπτεται από τη σχετική αξιολόγηση της ασπίδας, ε, κάτι το οποίο αναφέρεται ξεκάθαρα στα συμπεράσματα του Γενικού Εισαγγελέα. Όσον αφορά το P-Club, και τον ε, διαμεσολαβητή το γεγονός ότι δεν έχουμε εξετάσει λεπτομερό την διαδικασία είναι πράγματι μια ανησυχία για εμάς γιατί δεν έχουμε λάβει κάποιες καταγγελίες που μπορούν να γίνουν αποδεκτές ε, περιμένουμε κάποιες, δεν διαφημίζουμε κιόλας αλλά οπωσδήποτε αναμένουμε να έρθουν κάποιες ε, και αυτό θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί θα είναι η ευκαιρία να συζητήσουμε μεταξύ μας στους κεντρικούς φορείς της Ένωσης και στο προσωπικό του διαμεσολαβητή τις σχετικές διαδικασίες, γιατί οι διαδικασίες αυτές είναι απόρριτες. Και αυτό βεβαίως είναι μια ανησυχία, γιατί δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πλήρως τη λειτουργία του συστήματος, γιατί δεν ξέρουμε τις διαδικασίες, δεν ξέρουμε ποιε είναι και τι αποτελέσματα έχουν. Είναι ένα μαύρο κουτί. Οπότε, Τώρα, ε, επίσης υπάρχει ένα σχόλιο τη Κομισιόν ε, προς ε, εμά, αλλά δεν αφορά την Επιτροπή σα, Όσον αφορά την έκθεση ε, είναι συστάσεις για τις οποίες δεν ξέρουμε ακόμα αν ακολουθούνται ή όχι. Και σαφώς θεωρούμε ότι ακόμα και οι βελτιώσεις που επιφέρει η ΦΙΖΑ δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως, γιατί βεβαίως οι εγγυήσεις αυτές δεν αφορούν κατοίκους είπα, και έχει υπάρξει μια διαδικασία για να ξανανοίξει η διαδικασία αυτή που θα αφορά και τους ε, επιλογής ε, όχι μόνο τα δεδομένα γύρω από αυτούς οπότε είναι ευαίσθητη νομοθεσία η οποία πρέπει να τροποποιηθεί και πρέπει να δούμε τι αντίκτυπο θα έχει Νομίζω ότι αναφέρθηκα, απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Ε. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας, ε, τα επιπλέον και βεβαίως ε, να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες, να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Κομισιόν για τις προσπάθειες που έκαναν να απαντήσουν στις ερωτήσεις αυτές όπως πρέπει και αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι ε, ε, σεβαστήκατε και το χρόνο. Ε, βλέπω ζητάνε δύο συναλυτολόγους. Σας παρακαλώ ένα λεπτό. Κυρία Ίνετφελτ, μην ανησυχείτε κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Κοιτάξτε. πάντα θα υπάρχουν διαφορές στην πολιτική και νομική εκτίμηση μιας κατάστασης, αλλά ακούγοντας τους συναδέλφους σας, ε, η συνάδελφος εδώ πέρα υπερασπίστηκε μεγάλο πάθος στο αμερικανικό σύστημα. Η σκέψη δηλαδή ότι η προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας είναι στα χέρια σας, θα σας πω, πραγματικά με κάνει να χέζομαι πάνω μου. Έχετε κάποιο άλλο σχόλιο? Ε, και φρύτω όταν ακούω Ευρωπαίους αξιωματούχους να υπερασπίζονται τις αμερικανικές πρακτικές ε, μαζικής παρακολούθησης ενώ θα έπρεπε να προσπαθείτε να τις ε, σταματήσετε. Και βλέπουμε εδώ πέρα και την άποψη στην υπόθεση ΣΡΕΜΠ ότι η συλλογή δεδομένων πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία. Και δεν ε, υπάρχει εξουσιοδότηση για την αποθήκευση των δεδομένων. Δεν μιλάμε μόνο για παρακολούθηση, αλλά και την αποθήκευση. Και το δικαστήριο επίσης το έχει ξεκαθαρίσει αυτό στην απόφαση για την διατήρηση των δεδομένων, ότι η διατήρηση από μόνη τη είναι ε, μεγάλη παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα και δεν μπορεί να γίνεται διακρίτω. Και επιπλέον η απόφαση ΣΡΕΜΠ επίση λέει ότι χρειάζεται αποτελεσματική δικαστική ε, προστασία για την διαγραφή των δεδομένων μας και η ασπίδα αυτή ιδιωτικότητας ε, ούτε κατά διάνοια δεν ε, πλησιάζει σε αυτό. Ακούσατε. Λόγια σταράτα και κριτική στις απαντήσεις που δώσατε. Λοιπόν, έχετε τώρα δικαίωμα να απαντήσετε. Ε, σύντομα όμως παρακαλώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί έχουμε ήδη ε, απαντήσει. Ε, θα το επαναλάβω. Επιθυμήσαμε κάποια στοιχεία του αμερικανικού συστήματος ε, που συμπληρώνονται και από συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την ασπίδα ιδιωτικότητας και σε αυτά βαστήκαμε για το έβριμα επάρκειας. Αυτό το οποίο αναφέρεται ας πούμε, και στην άρθρο 702 του Αμερικανικού νόμου ε, είναι αντικειμενικό γεγονός. Αν δεν συμφωνούμε σε αυτό ε, είναι άλλο ζήτημα. Και πράγματι συμφωνώ με την κυρία Ινιτφέλντ υπάρχει ζήτημα ερμηνείας ε, και αυτό ακριβώς ε, και εδώ πέρα τελειώνω για να απαντήσω και στην κυρία Ζίπελ το δικαστήριο το ευρωπαϊκό γι' αυτό είπα ότι ε, θα χρειαστεί ίσως να επανέλθουμε τις επόμενους μήνες και εβδομάδες το δικαστήριο θα αποφασίσει όχι μόνο για την υπόθεση ΣΡΕΜΠ αλλά και για την διατήρηση των δεδομένων ε, και για το πρόγραμμα μαζικής ε, συλλογής ε, δεδομένων από κάποια κράτη-μέλη ή προσεχώς πρώην κράτη-μέλη, το Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή. Και εκεί πέρα θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα όσον αφορά την σχέση κάποιων δραστηριοτήτων από κρατικές αρχές και των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας και θα ξεκαθαρίσει και τα κριτήρια που ισχύουν όχι μόνο για ξένες χώρες αλλά και για τα κρατη και οπωσδήποτε ε, είναι πολύ ευπρόσδεκτη αυτή η διευκρίνηση στη δουλειά μας. Ναι, ναι. Πάνω στην ώρα είμαστε λοιπόν. Ωραία, σας ευχαριστώ. Και πάλι Εύχομαι τα καλύτερα για το νέο έτος. Θα τα πούμε στο Ρασβούργο την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.